Dear colleagues, in case you didn't notice, we are starting the meeting and I would like to, before I welcome... Σας καλωσορίσω εδώ. Ήρθε μόλις ο Αντιπρόεδρος. Θα ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά. Αποδοχή της ημερήσιας διάταξης. Έχει έρθει μια πρόταση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μετά από την συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς από τις 11 παρατέταρτο μέχρι τις 11.30 θα ακούσουμε τον Γκίγκολτ και μετά μέχρι τις 12 και τέταρτο θα ακούσουμε την, τις ψηφοφορίες και για την έκθεση Μπρέσο. Δεν υπάρχουν διαφωνίες. Η μερίσια διάταξη γίνεται δεκτή λοιπόν. Μία ανακοίνωση μόνο ήθελα να κάνω όταν Κρέντα έχει προταθεί σαν εισηγητής από το ΕΛΚΑ για την έκθεση της ΛΥΜΠΕ για το 2000, ε, την εφαρμογή της χάρτας για το 2014. Στο σημείο 4, έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων. Σεπτεμβρίου και 21 και 22 Σεπτεμβρίου είναι διαθέσιμα τα πρακτικά, θα θεωρηθούν αποδεκτά αν τυχόν δεν υπάρξει αντίρρηση κατατεθειμένη μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Περνάω λοιπόν στο επόμενο θέμα τώρα της ημερησίας ανταλλαγή απόψεων με τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Φραντ Τίμερμαντς. Στην αρχή ήταν υπεύθυνο για την καλύτερη διαχείριση, διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου και τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τώρα είναι υπεύθυνο για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ευρώπη και σίγουρα για τα θέματα που έχουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε. Συνεπώς του ευχόμεθα κάθε επιτυχία και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να εξηγήσω πού βρισκόμαστε τώρα καταρχάς το θέμα της διαφάνειας μετά από τη νέα μας πρωτοβουλία και πού ε, ελπίζουμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Την 1η Δεκεμβρίου οι Επίτροποι, τα γραφεία τους και η Γενική Διευθυντή συναντώνται μόνο με καταγεγραμμένους ε, λόμπιστ και δημοσιευμένους στα Μητρώα και στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν 2.400 ε, εκφραστές συμφερόντων υπέγραψαν το Μητρό από την 1η Δεκεμβρίου του 2014. Ε, μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, Goldman Sachs, Gazprom, HSBC, Coca-Cola, Heineken, όλα αυτά τα καλά παιδάκια. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα δεσμευτικό σύστημα, γιατί αν κάποιος δεν είναι στο Μητρό δεν μπορεί να συναντηθεί με αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι απλό. Οι επαφές με τους εμπλεκομένους κάθε φορά και τους ενδιαφερομένους είναι βασικό κομμάτι της διαδικασίας και όχι μόνο για μας αλλά για το σύνολο της Επιτροπής. Είναι απαραίτητο να μαζεύει κανείς όλες τις απόψεις για να καταλήξει σε κάποιες σωστές αποφάσεις και είναι απαραίτητο να δούμε πώς και ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει τις αποφάσεις που παίρνουμε ή που θέλουμε να πάρουμε. Αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις μας. Τα ίδια επίπεδα διαφάνειας για τα lobbying θα πρέπει να ισχύσουν και για τα τρία θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στη νομική διαδικασία, στην ομοθετική συγγνώμη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς κάναμε και μια πρώτα πρόταση για την διοργανική συμφωνία κοινού μητρώου που να καλύπτει και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτό. Και μάλιστα θα το αναδιοργανώσουμε χρονικά για να επιτρέψουμε να τεθεί ε, σε λειτουργία πρώτα η διοργανική συμφωνία για την καλύτερη διακυβέρνηση. Θα ξεκινήσουμε σύντομα και μια δημόσια διαβούλευση, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά τα οποία ακούσατε στην τελευταία σας δημόσια ακρόαση. Όπως επίσης και λαμβάνοντας υπόψη την εργασία του Sven Giegold. Υπάρχουν και μια ολόκληρη άλλη σειρά αλλαγών. Βελτιώσαμε τους κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες διαβουλεύσεις θα διαβουλευόμεθα πλέον και σε σχέση με τις κατεξουσιοδότης συμπράξεις και τις δευτερεύουσες νομοθετικές αποφάσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και μέσω του, του Δημοσίου Μητρώου ε, των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων. Προετοιμάζουμε κάποιες περαιτέρω αλλαγές για να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και το υπόλογο των συγκεκριμένων ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν διαδικασίες υποχρεωτικές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έτσι ώστε οι εκπρόσωποι συγκεκριμένων συμφερόντων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά να καταγράφονται και στο Μητρό Διαφάνειας. Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης της διαφάνειας και στην ομοθετική διαδικασία και για να πετύχουμε το στόχο αυτό στην πρόταση για την νέα διοργανική συμφωνία για καλύτερη νομοθεσία, προσκαλέσαμε και τα υπόλοιπα όργανα να δουν ακριβώς ποια είναι τα δικά τους επίπεδα διαφάνειας σε σχέση με τις ε, ε, νομοθετικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων μεταξύ των οργάνων. Θα υποστηρίξουμε και τις προσπάθειες από την επερχόμενη Ολλανδική Προεδρία, έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση ε, στα διάφορα μητρώα και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και με τους δύο συνομοθέτες γι' αυτό. Σύντομα τώρα για τη διαφάνεια στην εμπορική πολιτική, ιδιαίτερα σε σχέση με το TTIP. Όλοι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η συζήτηση για το TTIP μερικές φορές έχει γίνει επί τη βάση συναισθημάτων περισσότερο παρά γεγονότων. Ως εκ τούτου, έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαφάνεια που θα μας βοηθήσει να ξεχωρίσουμε τα πραγματικά γεγονότα σε σχέση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Βελτιώσαμε την κατάσταση, βελτιώσαμε το επίπεδο διαφάνειας και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την αμοιβαία κατανόηση και την αμοιβαία αντίληψη για τις διαπραγματεύσεις αυτές στο σύνολο της Ένωσης, λειτουργώντας με τον πλέον διαφανή και ορατό τρόπο. Δημοσιεύουμε τακτικά επεξηγηματικά μνημόνια Δημοσιεύουμε επίσης ε, νομικές πράξεις ε, για όλους τους τομείς της διαπραγμάτευσης. Έχουμε διευρύνει την πρόσβαση των Ευρωβουλευτών στα κείμενα πλευριορισμένης κυκλοφορίας, τα εμπιστευτικά έγγραφα και ξέρετε για τις αίθουσες ανάγνωσης κτλ. Οι προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις είναι θα έλεγα κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για σας, τα λεγόμενα consolidated text. Η Επίτροπος Μάλστρομ πάνω σε αυτό βρίσκεται σε επαφή με τον πρόεδρο της ΣΥΝΤΑ, τον κύριο Λάγκε, έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η πρόσβαση ε, των Ευρωβουλευτών στα έγγραφα αυτά τα σχετικά με το TTIP. Λοιπόν, είναι βασική η διαφάνεια για την σχέση μας, είναι όμως και βασική για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού. Η μυστικότητα γεννά τη μυθολογία και η μυθολογία γεννά αποστροφή προς την πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Yeah, you, can do it, no? Ναι, βεβαίως, μπορείτε να χειροκροτήσετε. But, yeah, now, dear colleagues, we, we συνάδελφοι. Θα ξεκινήσει η συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο και κατόπιν έχουμε 45 λεπτά χωρίς τον Αντιπρόεδρο με τον Σφεν Κίκολτ. Αν έχετε λοιπόν κάποιες δηλώσεις να κάνετε, αφήστε τις για το δεύτερο τμήμα. Έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο ομιλητών, ε, ενός είναι εδώ ο Αντιπρόεδρος και έχουμε χρόνο μέχρι τις 11 παρατέταρτο. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον εισηγητή. Καλώς ορίσατε. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι βεβαίως σας καλωσορίζουμε. Έχουμε κάνει κινήσεις και βήματα για περισσότερη διαφάνεια. Έχουμε δεσμευθεί σε θέματα ομάδων εμπειρογνωμόνων, αλλά και όσον αφορά τα διάφορα κείμενα που αφορούν τις ε, εμπορικές συναλλαγές. Μπορείτε βεβαίως να σχολιάσετε πρώτον το θέμα του μητρώου διαφάνειας. Αυτό θα γίνει δεσμευτικό, θα γίνει υποχρεωτικό. Ξέρετε ποια είναι η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς μιλήσατε για μια διαθεσμική συμφωνία. Μπορείτε να μας πείτε ξεκάθαρα πότε θα ξεκινήσει η διαβούλευση, πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε μια δική μας πρόταση, πότε θα έχουμε μια βάση για την οποία, την οποία θα στηριχτούμε για τη δική μας πρόταση. Μέχρι τώρα οι επίτροποι, από ό,τι μας είπατε, συναντώνται με εγγεγραμμένους στα Μητρώα εκφραστές ε, ομάδων συμφερόντων και θα ήθελα να μου πείτε αν και οι διαπραγματευτές υπόκεινται σε αυτήν την υποχρέωση. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί μέλη της Επιτροπής και συνεργάτες της οποίας οι οποίοι υπάγονται σε αυτούς τους κανόνες. Αυτό το μητρό διαφάνειας συμπεριλαμβάνει πολλά λανθασμένα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, το Μητρό, το αντίστοιχο στον Καναδά, έχει πολύ περισσότερους ελέγχους και ενημέρωση στοιχείων. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο και εσείς, μπορείτε να δεσμευτείτε εδώ ότι θα ελέγξετε πραγματικά την ακρίβεια των στοιχείων που συμπεριλαμβάνει αυτό το Μητρό. Τέλος, θέλω να αναφερθώ και στην ακαιρεότητα. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα μετά τις προτάσεις της διαμεσολαβήτριας, της συνηγόρου για βελτίωση και δεύτερον θεωρείται ότι αυτοί οι οποίοι ενημερώνουν την κοινή γνώμη ή οι whistleblowers μπορούν να προστατεύονται. Βλέπετε εδώ κάποιο τρόπο, μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα εργαστείτε για μια καλύτερη οδηγία όσον αφορά την προστασία αυτών των ανθρώπων. Και προτιμάτε όλες τις ερωτήσεις πριν να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, χαιρετίζουμε τον Αντιπρόεδρο. Βεβαίως δεν θα ε, θέσω την ίδια ερώτηση που έθεσα και χτες. Ε, ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις σχετικές. Η πρώτη είναι ένα ερώτημα, ένα ερωτηματικό. Τι συνέβη από απόψεως ε, διαφάνειας ε, με τις αντιπροσωπείες εάν ένα κράτος μέλος ε, προσπαθεί να σας επηρεάσει οι ομάδες, οργανισμοί ενός κράτους μέλους. Αυτό αποτελεί μέρος του Μητρώου ή όχι. Ή μια τρίτη χώρα ίσως, όχι μόνο μια χώρα μέλος. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη αφορά επίσης τη διαφάνεια Είμαι ο εισηγητής για το ECI και θα ήθελα να ξέρω αν η απόφαση λήφθηκε νομίζω με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, ε, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι γίνεται με άλλες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής ηθαγένειας και θα ήθελα να ξέρω αν το έγγραφο θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο για μας, προσβάσιμο για να δούμε με ποιο τρόπο λήφθηκε αυτή η απόφαση. Πρόκειται για το άρθρο 7 σχετικά με την Ουγγαρία. Να ξέρουμε από την, για το μέλλον, ε, για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες πολιτών, πώς λήφθηκε αυτή η απόφαση για να μπορέσουμε να ξέρουμε πώς κανείς φτάνει στο τέλος με ευκολία. Μπάρμπαρα Σπινέλη. Καλημέρα σας Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή την οποία κάνατε, το έτοιμά μου. Βλέποντας ότι οι αρμοδιότητές σας είναι πραγματικά τεράστιες. Περιλαμβάνουν και κάποια θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν ως ε, εισηγήτρια για την εφαρμογή ε, της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η ερώτηση την οποία θα ήθελα να θέσω έχει σχέση με αυτές τις τρομερές ε, τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τινησία, το Μαλί και το Παρίσι. Αυτό το οποίο με έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα στην αντίδραση της γαλλικής κυβέρνησης ήταν μια ιδέα όχι τόσο το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, το οποίο είναι δυσάρεστο αλλά είναι κατανοητό, αλλά η αναστολή εφαρμογής ε, της μεταβατικής ρήτρας 15, δηλαδή προσωρινή διακοπή της ελευθερίας κινητικότητας στο εσωτερικό του, Στέντεν, Σέγγεν που περιλαμβάνει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι ταυτόχρονα το Παρίσι είχε υιοθετήσει πολύ πρόσφατα έναν νόμο για τις ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός. Βλέποντας την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα δικαιώματα που καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στις προβλέψεις της Χάρτας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν το θέμα αυτό με την επίκληση της συγκεκριμένης ρήτρα είναι κάτι το οποίο θίγει άμεσα το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι στην ουσία σημαίνει ε, το να μιλάμε συνεχώς για κατάσταση πολέμου, για πιθανές συνταγματικές αλλαγές οφειλόμενες στο καθεστώς αυτό πολέμου. Μιλάμε για ένα νέο καθεστώς ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο λειτουργεί διαταρακτικά σε σχέση με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιολάινεν uh, για τους σοσιαλιστές. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητέ Φραντ, δεν είναι τυχαίο το ότι εδώ ζητάμε πολλά μέτρα για περισσότερη διαφάνεια και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Θα ήθελα να ζητήσω και εγώ πώς μπορεί αυτό το μητρό να συμπληρωθεί, να ολοκληρωθεί για την νομοθετική πράξη, πώς το, πώς το βλέπετε, πώς θα γίνει ολοκληρωμένο και δεσμευτικό αυτό το μητρό. Έχω και μία ερώτηση που αφορά την ε, σύγκρουση τα αντικρουόμενα συμφέροντα και με τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους συνεργάτες, μια επιτροπή τελικά και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το εργαλείο. Άκουσα 18 μήνες, 3 χρόνια. Θα πρέπει σίγουρα να επιστευτεί η διαδικασία. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην e-δημόκραση, ηλεκτρονική δημοκρατία, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, το e-voting. Σήμερα βλέπουμε ότι οι νέοι είναι στραμμένοι προς την ψηφιακή οικονομία και θα ήθελα να μου πείτε ο συνάδελφος Brooks, ε, δεν σας μίλησε για το Brexit. Θα το αναφέρω λοιπόν εγώ. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις θεσμικές συνέπειες ε, μιας ε, τέτοιας εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας και έχω την εντύπωση ότι καμία από τις ε, τέσσερις αν θέλετε ερωτήσεις που τίθενται δεν θα έχουν τελικά καθοριστική σημασία για το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δείξουμε μαλακή στάση, γιατί το αν θα μείνει ή αν θα φύγει η Μεγάλη Βρετανία σίγουρα θα εξαρτηθεί από άλλα πράγματα. Πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω. Πολλές ερωτήσεις θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ. Σχετικά με τον χρόνο για το Μητρό Διαφάνειας. Αυτό το οποίο κάναμε ε, είναι δεδομένου τη σχέση με το, με το Μητρό Διαφάνειας, ανάμεσα στο Μητρό Διαφάνειας και στην Διοργανική Συμφωνία για την Βελτίωση της Νομαθίας, θα, ε, για να, πριν από το τέλος του χρόνου να καταλήξουμε σχετικά με την διοργανή συνεργασία, διότι υπάρχουν στοιχεία ευξημένη διαφάνεια σε αυτή τη διοργανική συμφωνία και να θεωρήσουμε τη συμφωνία αυτή ως σημείο εκκίνησης και να έχουμε μια δημόσια διαβούλευση του χρόνου το συντομότερο δυνατόν και βάσει της δημόσιας διαβούλευσης να οριστικοποιήσουμε μια πρόταση για μια συμφωνία διοργανική για τη διαφάνεια για το μητρό της διαφάνειας. Ελπίζω να μπορέσουμε, και αυτό είναι μια απάντηση στην New ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο διαφάνειας το συμπεφωνημένο ανάμεσα στα όργανα, σε μια συμφωνία διοργανική, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να δημιουργήσουμε δεσμευτική νομοθεσία, αλλά ίσως χρειαστεί αυτό να γίνει οπωσδήποτε, αλλά πρέπει να δούμε πόσο μακριά θα μπορέσουμε να φτάσουμε με μια συμφωνία διοργανική. Θα ήθελα τα πράγματα να γίνουν με αυτή τη σειρά. Βεβαίως, δεν θα διστάσω να προχωρήσω με νομοθετική ε, εργασία, αλλά αυτό ξέρουμε ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και θα είναι πιο δύσκολο να γίνει αυτό και να συμφωνηθεί με το Συμβούλιο από ότι να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε με μια διοργανική συμφωνία. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό σχετικά με τη στιγμή, με το χρόνο όπου θα δημοσιοποιήσουμε τις αποφάσεις ε, που, θα, που λαμβάνονται το Δεκέμβριο ε, για την ε, καταγραφή, την καταχώρηση όλων των συναντήσεων. Βεβαίως, οι κριτικές μερικών από εσά αλλά και από έξω ήταν βεβαίως πολύ καλό πρώτο βήμα, αλλά θέλουμε όλοι να περιληφθούν στο Μητρό όσοι εργάζονται στην Επιτροπή για θέματα πολιτικής. Δεν συμφωνώ με αυτή τη θέση, διαφωνώ επειδή θα ήθελα αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις να είναι σε αυτόν τον κατάλογο και οι αξιωματούχοι ε, δεν είναι πάντοτε αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις είναι αυτοί που οριστικοποιούν τις αποφάσεις και αυτοί που τελικά έχουν την ευθύνη για αποφάσεις αυτές και θα πρέπει να είμαστε σαφείς για το ποιους συναντούν. Ξέρω ότι θα είναι μια συνεχιζόμενη συζήτηση, θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Είμαι ανοιχτό για αυτή τη συζήτηση και δεν, δεν θέλω να είμαι ιδεολόγος, θέλω να, είμαι, ε, να κάνουμε πρακτικά βήματα, να έχουμε μια συζήτηση για το πού θέλουμε να σταματήσει αυτή η διαδικασία διότι σε κάποια στιγμή, σε οποιαδήποτε οργάνωση, οργανισμό, το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι, νομίζω, θα πρέπει να προστατευτούν από την δημόσιο έλεγχο, διότι δεν είναι όλοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Χρειάζεται μια ισορροπία να επιτευχθεί ανάμεσα στην ανάγκη διαφάνειας για αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και την ευθύνη που έχουμε ως επικεφαλής ενός οργανισμού, να προστατεύσουμε επίσης την ακαιρεότητα και μέχρι ενός ορισμένου σημείου την ιδιωτικότητα αυτών που εργάζονται. Πρέπει να έχουμε ε, μια, μια ισορροπία. Ε, αλλά είμαι ανοιχτό ε, για συζήτηση. Δεν, δεν είμαι δεγματικός. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή με άλλους οργανώσεις, την Transparency International που έχει πολύ πείρα στον τομέα. Προσπαθώ να βρω τη σωστή ισορροπία εδώ. Και Ξέρω ότι ο Σβέν Γκίγκολντ έχει κάνει πάρα πολύ καλή εργασία και έχει τοποθετήσει σχετικά με το θέμα αυτό. Αλλά όπως είπα, ο Σβέν Γκίγκολτ και εμείς και εγώ δεν διαφωνούμε για το θέμα αυτό, αλλά δεν πρέπει μόνο να κατηγορούμε την Κομισιόν θα είναι επίση ένα μεγάλο βήμα προ τα μπρο αν τα μέλη του Κοινοβολίου συμφωνούν για πλήρη διαφάνεια και δεχθούν να καταχωρίζονται όλες οι συναντήσεις τους. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσά το πράττουν, το θέλουν, γιατί να μην το κάνουμε πιο επίσημο, να μην το ε, τυποποιήσουμε Ξέρω ότι ένας από εσά σε μια συνάντηση που είχα στη συζήτηση είπε ότι είμαστε επιφυλακτικοί. Είμαι επιφυλακτικός. Αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά ίσως ε, είσαστε επιφυλακτικοί, ίσως επειδή είστε εκλεγμένοι. Τότε είναι μεγαλύτερη η ευθύνη σας. Θα πρέπει να διευκρινίσετε στους ψηφοσόρους σας ε, τι κάνετε, ποιους συναντάτε, για το τι μιλάτε. Ναι, ναι, καταλαβαίνω, αλλά μπορείτε να έχετε και τις δύο προσεγγίσεις στο θέμα αυτό και δεν βλέπω γιατί εάν ένα θεσμό ως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Κομισιό να είναι στο δυνατόν πιο διαφανής και να καινοτομεί και να προχωρήσει ο δρόμο αυτό ενώ η Επιτροπή μπορεί να πει στο Κοινοβούλιο γιατί να μην το κάνουμε από κοινού και να μην ακολουθείτε κι εσείς το παραδειγμά μας και να κάνετε το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθούσε ε, να, διαμορφώσουμε την δημόσια εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι ο κάθε επίτροπος, ε, το κάθε γραφείο επιτρόπου, ο κάθε γενικός διευθυντής ε, είναι υπεύθυνος για την ποιότητα. Και είναι μια διαδικασία εκμάθησης την οποία έχουμε εδώ και ένα χρόνο βεβαίως. Μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα και σας καλώ να μας δώσετε ορισμένε ενδείξεις για το πού θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αναφέρατε το καναδικό παράδειγμα θα ήταν καλό το παράδειγμα αυτό. Είμαι διατεθειμένος να ζητήσω από την ομάδα μου να το εξετάσει και να μας δώσει μερικές συμβουλές για το πώς να βελτιώσουμε τα πράγματα, αλλά το είπα ρητά σε όλους τους συναδέλφους μου ότι δεν μπορείτε ε, να θεωρήσετε άλλους υπεύθυνους. Εσείς είστε υπεύθυνοι ε, εσείς πρέπει να κάνετε τα πράγματα σωστά και εσείς πρέπει να λογοδοτείτε και θα θεωρηθείτε υπεύθυνοι προς τον εξωτερικό κόσμο εάν δεν κάνετε σωστά τα πράγματα. Αλλά βεβαίως αυτό δεν είναι τέλεια η κατάσταση, πρέπει να μαθαίνουμε ημένα από τους ΔΕ και να βλέπουμε τα παραδείγματα αυτών που κάνουν καλύτερη εργασία. Σχετικά με το revolving doors, ε, αυτήν ε, την ε, αλλαγή συμφερόντων ορισμένων που έχουν ηθήνουσες θέσεις και χρησιμοποιούν για να κάνουν άλλες δουλειές. Έχουμε την περίοδο με τη μεταβατική, το cooling off, το άρθρο 2, 45, μας δεσμεύει και θα πρέπει να έχουν ε, κατάλληλη συμπεριφορά αφού ε, σταματήσανε να έχουν ένα λειτουργήμα και σταματήσανε να έχουν αμοιβέ ε, και προνόμια. Δεν υπάρχει όριο σε αυτή την αρχή. Η διάρκεια της υποχρέωσης κοινοποίηση στην Επιτροπή ε, είναι χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη. Η περίοδος των 18 μηνών είναι αρκετή εφόσον επιτρέπει στην πράξη να χαλαρώσουν οι σχέσεις ανάμεσα έναν πρώην επίτροπο και το θεσμικό όργανο. Νομίζω ότι η παράταση που προτάθηκε θα είναι και μιλάει ο Επίτροπος που είναι υπεύθυνο για καλύτερη νομοθεσία, ότι δεν είναι απαραίτητη ε, κουρατικά αυτή η παράταση και δεν θα έχει περαιτέρω προστιθέμενη αξία και δεν είμαι υπέρ της παράτασης αυτής της μεταβατικής περίοδου. Σχετικά με τους whistleblowers, τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ε, θα μας... Ε, θα θα πρέπει το προσωπικό να μπορεί ε, να καταγγέλει ανάρμοστη συμπεριφορά, να πληροφορεί για ανάρμοστη συμπεριφορά ε, και όσοι θα το πράττουν δεν πρέπει να τιμωρούνται, αλλά να προστατεύονται δεόντως κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας. Δεν προβλέπουμε μια οδηγία όπως ε, πρότεινε ο Σβεν Ε, για στοιχεία νομοθεσίας έχουμε κανόνες σχετικά με τους whistleblowers. Ξέρω ότι το συζητάτε αυτό σχετικά με το σχέδιο νομοθεσίας για τα εμπορικά μυστικά και απόρριτα και παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων δεν έχουν υποχρέωση να ε, καταχωρίζονται το είπα στον κύριο Σέπλιν, σχετικά με το ECI και το άρθρο τα κόσα πήραμε ε, την απόφαση την ε, τελευταία εβδομάδα. Αν δεν είχαμε λάβει την απόφαση εκείνη τη εβδομάδα θα είχαμε παραβιάσει την περίοδο των τριών μηνών όπου έπρεπε να λάβουμε απόφαση. Συνεπώς είμαι υπερήφανος ε, βεβαίως ήταν την τελευταία εβδομάδα, αυτό σημαίνει ότι δεν βιαστήκαμε και πάλι η θέση της Επιτροπής ε, δεν λέει τίποτα για το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας όπως θα καταλάβατε. Είναι μια νομική θέση που λαμβάνουμε όταν, όταν λαμβάνουν την πρωτοβουλία οι πολίτες. Πρέπει να δούμε αν αυτό συμφωνεί με τους κανόνες και θα πρέπει να εξετάσουμε το γεγονός εάν είναι για ένα θέμα το οποίο απαιτεί μια νομική πράξη. Με αυτή την έννοια δεν είχαμε αντίρρηση σχετικά με την πρωτοβουλία, με την ECI, αλλά όπως είπε ο Επίτροπος εχθές στη συζήτηση για την Ουγγαρία, η Επιτροπή δεν έχει κανένα λόγο να αρχίσει η διαδικασία του άρθρου 7 κατά της Ουγγαρίας, εάν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος, βάσιμος λόγος γι' αυτό, θα το πράξουμε και δεν χρειαζόμαστε ECI για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Ε, σχετικά για την ECI δεν μπορεί ε, να υποχρεώσει την Κομισιόν για το άρθρο 7, διότι το άρθρο 7 έχει μια σαφή πρόθεση, μια σαφή διαδικασία και θα πρέπει να κρίνει η Επιτροπή αν θα την ακολουθήσει ή όχι. Κατ' ουδένα τρόπο δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας πολιτών. Θα είμαι πιο σύντομος τώρα. Η κυρία Σπινέλη ρώτησε, έθεσε μια πολύ περίπλοκη ερώτηση. Όπως γνωρίζετε, στις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ζητήθηκε μια νομοδότηση της Επιτροπής και δόθηκε και στη Γαλλία. Θα συμφωνήσετε μαζί μου να σας δώσω μια γραπτή απάντηση γιατί πρόκειται για θέματα νομικά περίπλοκα και δεν θα ήθελα να κάνω λάθη εδώ απαντώντας πρόχειρα. Λοιπόν, αν δεν σας πειράζει, ε, θα σας δώσω μια γραπτή απάντηση. Ευχαρίστως, λέει η κυρία Σπινέλη. Τώρα για το e-voting και το Brexit για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, για την ευρωπαϊκή, συγγνώμη, ευρωπαϊκού τύπου ψηφοφορία. Προφανώς και θα ήμουν υπέρ, ε, αλλά δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές στον εκλογικό πολιτισμό της κάθε χώρας σε σχέση με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, να συγκρίνει κανείς με την, την Εστονία με τη Γαλλία ή με την Ολλανδία. Στην Εστονία, ας πούμε, οι πολίτες το χρησιμοποιούν με τον πολύ, ε, ε, πολύ πιο εύκολα από ό,τι σε άλλες χώρες τα ιατρικά τους στοιχεία κτλ. Λοιπόν, ε, αν προσπαθήσουμε να έχουμε λοιπόν ένα κοινό ευρωπαϊκό έδαφος σε σχέση με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, απαιτείται χρόνος. Και δεν μπορούμε παρά να σεβόμαστε τις διαφορές ανάμεσα στις διάφορες χώρες, αλλά το μέλλον βρίσκεται εκεί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και τέλος για τον Brexit. Θα ήταν άδικο για τον κύριο Σέπλιν να απαντήσω στην ερώτησή σας κύριε Λάιον έχοντας πει χθε στον κύριο Σόπλινγκ ότι στην παρούσα φάση δεν θα ήταν ιδιαίτερα σοφό για μένα να σχολιάσω τα τέσσερα σημεία τα οποία έθεσε στην ομιλία του ο κύριος Κάμερον. Συνάδελφοι, αν θέλετε να δώσετε την δυνατότητα στον Αντιπρόεδρο να δώσει κάποιες απαντήσεις, όχι, δύο, όχι πάνω από δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Γιαζόφσκι, ε, ομάδα των συντηρητικών. Ε, Panie Komisarzu, bardzo dziękuję za, e, za te deklaracje i działania. Ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας σχετικά με τη διαφάνεια. Δύο θέματα θέλω να ρωτήσω. Καταρχάς να συμφωνήσω με τον κύριο Σόφλε. Και εγώ πιστεύω ότι το θέμα το οποίο έθεσε η Ουγγαρία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με τη συγκεκριμένη αυτή ρύθμιση που δίνει την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει από τα κάτω μια δυνατότητα διαδικασίας νομοθετικών ρυθμίσεων. Αυτό ήταν ένα σχόλιο. Τώρα, πώς αξιολογείται ε, την πρόοδο των διοργανικών, τι μάλλον των διαπραγματεύσεων για τη διοργανική συμφωνία. Η κυρία Μπρέσο και ο κύριος Μπροκ σε μια ανακοίνωσή τους αναφέρονται ασκώντας κριτική στην πρακτική ε, υπογραφής, ε, ολοκλήρωσης μάλλον ε, συζητήσεων για συμφωνίες μετά το τέλος της πρώτης ανάγνωσης. Η κυρία Μπρέσο και ο κύριος Μπρόκ θεωρούν ότι αυτή σαν πρακτική δεν είναι σωστή και αγνοεί ουσιαστικά τον ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποια είναι η άποψη λοιπόν της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σύναψη αυτή ε, των συμφωνιών αμέσως μετά την πρώτη ανάγνωση. Θα ήθελα τι απαντήσει σας. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ Επίτροπο και εγώ θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση η οποία έχει σχέση με τον κύριο Γκίκολτ για το Μητρό Διαφάνειας. Είπατε εσείς τι βήματα έχουν γίνει από πλευρά σας, είπατε επίσης και τι βήματα σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον και με τα οποία συμφωνούμε αλλά υπάρχει και η δυνατότητα της προσωπικής ε, πρόσβασης σε την δυνατότητα αμφισβήτησης μιας απόφασης. Το θέμα είναι να μην μείνουμε στη ρητορία. Έχουμε τον κόσμο ο οποίος είναι απαραίτητος για να φέρει εις πέρας ε, τις ε, διαδικασίες αυτές με σωστό τρόπο. Μπορείτε να μας πείτε ότι πέρα από τις αποφάσεις σε επίπεδο πρακτικής, αυτά τα οποία ε, προβλέπεται μπορούν να λειτουργήσουν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, σε σχέση με την λεγόμενη αυτή διαδικασία των περιστρεφωμένων θυρών. Ας υποθέσουμε ότι ένας υπουργός σε μια χώρα γίνεται επίτροπος Και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, εν πάση περιπτώσει. Αυτό συμβαίνει. Ξέρετε ότι ο, ο κύριος Κανιέτε, ο επίτροπος Κανιέτε ήταν υπουργό προηγούμενη κυβέρνηση Γεωργίας και μετά παρετήθηκε ήταν επιχειρηματίας φυσικά, ήταν επιχειρηματίας με συμφέροντα διακήρυσης ε, ε, πολλών, ε, σε πολλούς τομείς στην Ισπανία και αυτό δημιουργεί μια σύγκρουση συμφερόντων. Θα ήθελα να μάθω ε, τι σκέφτεστε γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε να κάνουμε με μια πραγματική υπόθεση. Δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Thank you uh, very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φάβιο Καστάτα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Τίμερμαν, στον ευχαριστώ που είναι μαζί μας για να συζητήσουμε. Επιστρέφω στο θέμα του Μητρώου Διαφανείας. Μας μιλήσατε κυρίως για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο, αλλά έχει σημασία και ποιες είναι οι θέσεις που ακούγονται στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πιέσουμε το Συμβούλιο έτσι ώστε να υιοθετήσει κάποιες από τις προτάσεις που κάνατε σήμερα, τις τόσο θετικές θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι στο μέλλον τουλάχιστον και πέρα από τη διοργανική συμφωνία θα πρέπει να είμαστε ε, πιο φιλόδοξοι σε σχέση με τον κανονισμό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη νομική βάση που βρίσκεται από πίσω και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην αποτελεσματικότητα των αποφασεών μας για την διαφάνεια τώρα της νομοθετικής διαδικασίας, των νομοθετικών διαδικασιών. Έχει μεγάλη σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση να είμαστε ε, βέβαιοι για τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα η οποία θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα έγγραφα, τα οποία πολλά από αυτά σήμερα δεν είναι διαθέσιμα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και καθορίζουν το νομοθετικό ήτερ των αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε εκφράσεις θέσεων, αλλά σε συγκεκριμένες ενέργειες. Για το TTIP, εσείς ε, μιλήσατε για την ε, ανάγκη βελτίωσης του τρόπου με το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξηγηθεί σωστά. Εγώ άκουσα κάποιες κάποια τριαμβευτικά σχόλια <clears throat> για την βελτίωση των τρόπων με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση. Και μάλιστα είχαμε ακούσει ότι και το θέμα το οποίο συζητήθηκε στα πλαίσια του TTIP της ιδιωτικής διαιτησίας είναι κάτι το οποίο έχουμε, στο οποίο έχουμε ήδη υπερισχύσει. Ε, το θέμα είναι ότι στην ουσία εσείς προτείνατε ε, μια διαφορετική αντίληψη για την ιδιωτική διαιτησία. Δεν την έχετε πετύχει ακόμα. Οπότε λοιπόν εφόσον πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, πρέπει να υπάρξει διαφάνεια για 360 μοίρες και όχι να διαλέγετε επιλεκτικά κάποια θετικά στοιχεία και αυτά να τα υπογραμμίζετε. Τέλος, <clears throat> ένα συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο συνδέεται με το άρθρο 42 της εκθέσεως του κυρίου Γκίγκολντ για την περίοδο cooling off σε σχέση με, τα, με τη σύγκρουση συμφερόντων. Ίσως, και το λέω εδώ και σαν μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, και στη συγκεκριμένη πρόταση οδηγίας και στις διαδοχικές οδηγίες να συμπεριλάβουμε επίσης και κάποιες, ε, κάποιες θέσεις, εν πάση περιπτώσει, τις οποίες ε, δημιουργούμε, ε, του ειδικού εκπροσώπου, του ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι υπάρχει ας πούμε η θέση του κυρίου Λεόν, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα της ε, νότιας περιοχής της Μεσογείου, ο οποίος διορίστηκε σε μία άλλη θέση των Ηνωμένων Εθνών και αμέσως μετά διορίστηκε πρόεδρος της ε, Διπλωματικής Ακαδημίας ε, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στις διαπραγματεύσεις στη Λίβη και έχει κάνει τα Ηνωμένα Έθνη να χάσουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αξιοπιστίας το οποίο είχαν το εσωτερικό των διαπραγματεύσεων αυτών έχει υπονομεύσει και τη θέση του ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις με την Λιβύη. Συνεπώς λοιπόν αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να διευρύνουμε την περίοδο αυτή την τριετή και στις θέσεις των ειδικών αντιπροσώπων. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα τους δώσουμε και μεγαλύτερη ελευθερία βέβαια σε σχέση με τους υπαλλήλους αυτούς καθεαυτούς της Ένωσης. Ο κύριος Κόμπετ. Ευχαριστώ. Δεν θα κάνω ερώτηση εγώ για το Brexit, το λεγόμενο Brexit. Πραγματεύσεις της Μεγάλης Βρετανίας που είμαι σίγουρη ότι φυσικά θα γίνουν με μεγάλη διαφάνεια, με ανοιχτό πνεύμα και ότι όλοι θα γνωρίζουμε ποιες είναι οι διάφορες προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις που βρίσκονται στο τραπέζι και συζητούνται μεταξύ Βρετανών και Συμβουλίου. Αυτό που θα ρωτήσω είναι πολύ συγκεκριμένο. Ένας φορέας, ένας οργανισμός, μια εταιρεία η οποία βρίσκεται σε αυτό το κοινό μητρό και παραβιάζει κανόνες μπορεί να βγει από αυτό το μητρό με μια ατομική απόφαση ενός θεσμού, ενός θεσμικού οργάνου ή δεν θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο εάν δεν υπάρξει συνένεση και συμφωνία των όλων των θεσμικών οργάνων. Πώς δηλαδή μπορεί να βγει μια εταιρεία ή ένας φορέας. Και αυτό όχι μόνο εάν παραβιάζονται οι κανόνες ή παρόμοια περίπτωση θα μπορούσε να προκύψει εάν μία επιχείρηση δεν συνεργάζεται. Δεν θα πρέπει να τους πούμε με κάποιο τρόπο ότι αφού δεν συνεργάζεστε μαζί μας, δεν θα συνεργαζόμαστε και εμείς μαζί σας και δεν θα υπάρχει από εκεί και πέρα καμία απολύτως στήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κ. Σόλτς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των εμπορικών συναλλαγών και της διαφάνειας. Βεβαίως εδώ προσπαθούμε να φτάσουμε σε μία επισημοποίηση αυτών των μητρώμων. Αλλά και ο κύριος Λάγκε όταν τοποθετήθηκε στην έκθεση Giggold αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Στο θέμα δηλαδή της, του μεγάλου αριθμού διαφόρων διαπραγματεύσεων, συζητήσεων οι οποίες γίνονται με δική μας εντολή σε πολλούς τομές. Παραδείγματο χάρη θέματα αγροτικά, θέματα οικονομικά, στα πλαίσια της ε, συμφωνίας TTIP. Και οι εντολές αυτές υπάρχουν, αναρωτιέμαι όμως αν όλα αυτά ενσωματώνονται σε αυτό το Μητρό ή εάν ουσιαστικά ρυθμίζονται από μία συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Είναι συγκεκριμένο, γνωρίζουμε ποιος διαπραγματεύεται πού και αν εντοπίζονται τα βήματα πρόοδου. Εμείς πού βρισκόμαστε αν θέλετε στα πλαίσια παραδείγματος χάρη των διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα με τρίτες χώρες ποιοι είναι οι φορείς, ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ποιος διαπραγματεύεται σε ποιο επίπεδο. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αυτό το Μητρό Διαφάνειας ενσωματώνεται στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες που ξέρουμε ότι λαμβάνουν χώρα. Και βεβαίως το θέμα της ε, περαιτέρω προόδου στην διοργανική συμφωνία έχει βεβαίως και αυτό κάπου τη σημασία του εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία ερώτηση από τον κύριο Σόπελ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι ο συνάδελφος ο οποίος μου έδωσε την ε, ερώτηση αυτή είναι στη Βενεζουέλα, παρατηρητής των εκλογών. Θα τη διαβάσω λοιπόν. μετά από έτοιμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλο, επιτέλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τις προτάσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμφωνία του 2003 για καλύτερη νομοθεσία. Και ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος έλαβε και την εντολή, είναι γνωστό. Σήμερα γνωρίζουμε επίσης ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΕΛΚ όσον αφορά αυτήν την διαπραγμάτευση και την αναθεώρηση. Ανεξαρτησία, σαφής κανόνες για τη διαφάνεια, έλεγχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων και των φορέων που λαμβάνουν χώρα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και βεβαίως να υπάρχει εδώ ίση μεταχείριση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει εδώ να βρίσκεται σε μια ίση θέση με το Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το ΕΛΚ συγκεκριμένα να γίνεται έλεγχος εντελεχής και βεβαίως να λαμβάνεται εδώ και να στηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Θα θέλαμε να ξέρουμε εάν λαμβάνονται υπόψη και οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι συνεργάζονται με την Επιτροπή, όχι μόνο δηλαδή οι συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν συμπεριλαμβάνονται σε, αυτές, σε αυτούς τους ελέγχους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για την πολιτική ομάδα του ΕΛΚ η εκτίμηση και του ετήσιου ε, κόστους. Θα θέλαμε να ξέρουμε πώς μπορούν να συνεχιστούν σε αυτό το πλαίσιο και οι διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, τι θεωρείται παράνομο και τι όχι και όσον αφορά τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης και αν αυτές ε, μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτές τις διαδικασίες και φαντάζομαι έχει ένα ερωτηματικό στο τέλος. Σας δίνω το λόγο κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήδη απήντησα στην ερώτηση σχετικά ε, με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, την ECI, αλλά καταλαβαίνω ε, την θέση σας ε, που είναι, ευθυγραμμίζεται με τη θέση του κ. Τσέπλιν. Σχετικά με την πρώτη ανάγνωση έκανα ένα λάθος σε προηγούμενη φάση, σε συνάντηση σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξέφρασα μια γνώμη για την πρώτη ανάγνωση και αμέσως είχα την αντίδραση του Κοινοβουλίου, σωστά, ότι δεν θα έπρεπε να ε, αναμειγνύομαι σε πράγματα που δεν με αφορούν, σε υποθέσεις που δεν με αφορούν, διότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει για το θέμα αυτό. Ε, παρόλο που θα ήθελα να επαναλάβω ε, τη θέση μου, είναι πειρασμός για μένα, δεν θα το πράξω σεβόμενος τις αρχές που είναι υπεύθυνε για να αποφασίσουν αν υπάρχει μια πρώτη διαδικασία συνδιαλλαγής ή όχι. Συνεπώς, Εάν όμως προσεγγίσετε το θέμα από την άποψη της διαφάνειας και καλύτερης νομοθέτησης και κάνετε μια γενική παρατήρηση χρησιμοποιώντας καμιά φορά ολόκληρο το φάσμα της λήψης αποφάσεων θα μπορούσε δυνητικά να δώσει καλύτερα αποτελέσματα από το να επιλέξει κανείς να πάει για συνδιαλλαγή στην πρώτη ανάγνωση. Νομίζω μπορώ να το πω χωρίς να προκαλώ οργή από την άλλη πλευρά. Και σχετικά με το μητρό διαφανείας και για να βελτιώσουμε την ποιότητα. Αυτή ήταν και πάλι η πρώτη ερώτηση. Έχουμε και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, έχουμε προσωπικό που εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό, γιατί δεν ζητούμε την γνώμη του προσωπικού και θα μπορούσαμε με βάση τη γνώμη αυτή να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα όταν είναι ουριάνεμη και θα δούμε σε τελευταίο στάδιο αν μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι μόνο το θέμα να αυξήσουμε το προσωπικό. Αυτή συνήθως σε κάθε διοίκηση είναι η συνήθις λύση, προσθέτουν άτομα στο προσωπικό. Δεν ξέρω αν ωφελεί. Θα ήθελα να είμαι σύντομος ε, για να δούμε πού είναι τα προβλήματα, πού είναι οι λήψεις, ε, προτού περάσουμε ε, σε άλλη κατεύθυνση. Και μετά από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί από εσά θέλουν να θέσουν ειδικά θέματα σχετικά με ειδικά άτομα. Όχι, όχι, δεν θα μπω σε ατομικές περιπτώσεις μαζί σας. Συζητούμε τις γενικές αρχές, αλλά δεν θα συζητήσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Νομίζω ότι οι διαδικασίες υπάρχουν, αν υπάρχει μια ατομική περίπτωση, αυτό θα έρθει στο φως αλλά και υπάρχουν διαδικασίες, αλλά εδώ θα συζητήσω συγκεκριμένες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι καμιά φορά υπάρχει ένα πολιτικό θέμα εκεί και δεν πρόκειται να αναφερθώ στις περιπτώσεις αυτές σε αυτή τη συνάντηση. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν για όλους, για όλους που εργάζονται στην Επιτροπή όλα τα τμήματα της Επιτροπής. Ο κύριος Καστάλντο ρώτησε εάν δεν πρέπει εκτός αυτών να νομοθετήσουμε για την, το Μητρό Διαφάνειας. Θα ήθελα να επαναλάβω Ας προσπαθήσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε διαμέσου μιας διοργανικής συμφωνίας. Αν δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα θα εξετάσουμε την δυνατότητα μιας νομοθεσίας για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Αλλά αυτή θα είναι η δεύτερη επιλογή μου. Η πρώτη επιλογή μου ως προς το επίπεδο διαφάνειας, ακόμα και των πρακτικών, θα πρότεινα να να, είναι αυτό, να γίνει αυτό ένα θέμα συζήτηση όταν συζητήσουμε την διοργανική συμφωνία, να δούμε μέχρι ποιου σημείου πρέπει να έχουμε διαφάνεια. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να συζητήσουν και τα τρία θεσμικά όργανα. Ο κύριος Καστάλντο ε, ζήτησε εξηγήσει, προσπαθώ να τις δώσω τώρα, μια εξήγηση ε, που μπορώ ε, να τον ρωτήσω τι γίνεται με την Ρώμα Προβίνσκα. Είπα, Ρώμα. Είχαμε την ίδια πάθος ε, για την ίδια ομάδα ποδοσφαίρου. Ο κύριος Κόμπερτ ρώτησε τι πρέπει να γίνει μετά την παραβίαση. Οι κανόνες είναι σαφείς στο Μητρόλο. Ίσως ε, δεν εάν ε, είναι ίσως αυτή η ερώτηση, αν ε, παραβιάσει κανείς τους κανόνες, διαγράφεται από το Μητρό, θέλετε να ρωτήσετε εάν ένα όργανο αποφασίσει να διαγράψει κάτι ή κάποιον από ένα μητρό, αυτό θα πρέπει να ισχύσει και για τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Ναι, νομίζω πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι δεν μπορείτε να λάβετε ως όργανο μία μονομερή απόφαση. Αυτό κάθε θεσμικό όργανο είναι ελεύθερο να το πράξει, αλλά νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση που θέλουμε να συζητήσουμε όταν θα έχουμε τη γενική συζήτηση για την προετοιμασία της διοργανικής συμφωνίας θα είναι να δούμε εάν αυτή η απόφαση από ένα όργανο θα προκαλέσει απόφαση από άλλα όργανα. Διότι νομίζω ότι υπάρχει εδώ κοινό συμφέρον. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό χωρίς να προκαταλαμβάνω την θέση που θα υιοθετήσω, καταλαβαίνω την λογική της συνεργασίας μεταξύ των τριών οργάνων, χωρίς βεβαίως να προκαταλαμβάνουμε το δικαίωμα του κάθε οργάνου να λαμβάνει μια τέτοια απόφαση. Αυτή θα ήταν η προσέγγιση μου στο θέμα αυτό. Σχετικά με την εντολή διαπραγμάτευσης. Θα ήθελα να είμαι σαφής απέναντι στον κύριο Σόλτς. Δεν υπάρχει καμιά διαπραγμάτευση στον κόσμο που να μην έχει ένα μέρος απορρίτου. Δεν μπορείτε να διαπραγματεύεστε μια διεθνή εμπορική συμφωνία με πλήρη διαφάνεια. Εκτός εάν όλα τα μέρη ζητήσουν πλήρη διαφάνεια. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Αν θέλετε να διαπραγματεύεστε επιτυχώς θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να συμβουλεύεστε αυτούς από τη δική σας πλευρά χωρίς η άλλη πλευρά να ξέρει τι συζητάτε με τους δικούς σας και προς τα πού το πάτε. Διότι δεν μπορείτε να διαπραγματεύεστε. Αν διαπραγματευτείτε με την άλλη πλευρά με απόρριτο τρόπο είναι καλό. Αλλά αν είναι ανοιχτή η δημόσια η θέση σας, δεν ε, θα επιτύχετε στη διαπραγμάτευση. Πρέπει να υπάρχει με ένα επίπεδο εμπιστοσύνης στο Συμβούλιο προτού ε, διαπραγματευτείτε. Θα πρέπει να δείξετε στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης το δίδιο επίπεδο διαφάνεια διότι τώρα υποχρεώνουμε τους Αμερικανούς να είναι πολύ πιο διαφανείς από ό,τι το επιθυμούν και υπάρχει κάποια επιτυχία, αλλά πλήρης διαφάνεια σε μια διαπραγμάτευση. Όποιος έχει ασχοληθεί με την πολιτική παραπάνω από μια μέρα ξέρει ότι αυτό είναι ανέφικτο για όλες τις διαπραγματεύσεις εμπορικές πολιτικές. Αν επιζητείτε ένα συμβιβασμό πρέπει να προστατεύσετε την θέση ε, των άλλων για να οδηγηθείτε σε ένα συμβιβασμό. Ή το μόνο που έχετε είναι να χάσετε και αυτή είναι η αρχή, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για περισσότερη διαφάνεια στην εντολή που δίδεται. Δεν το αμφισβητώ αυτό, δεν μπορείτε να ζητήσετε από το Συμβούλιο να είναι τελείως ανοιχτό με την εντολή, διότι ε, θα γνωστοποιήσει την διαπραγματευτική θέση πρωτού αρχίσει η διαπραγμάτευση. Και το τελικό μου σημείο για τον κύριο Σάπλιν. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα είπατε, αλλά νομίζω θα πρέπει να τα πείτε αυτά στον κύριο Φερχόφσταντ, διότι αυτός διαπραγματεύεται εκ μέρους του Κοινοβουλίου με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αλλά χωρίς ε, να προκαταλαμβάνω τη θέση του κυρίου Βερχόφστατ, τα στοιχεία που αναφέρετε είναι μέρος της διαπραγμάτευσης και ελπίζω να μπορείτε να βρείτε ένα συμβιβασμό για όλα αυτά τα στοιχεία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν πολλά προβλήματα ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Δεν νομίζω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα σας ξαναδούμε. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε καλό. Θα συνεχίσουμε με τον Σφεν τη συζήτηση. question, Δεν έχω ερώτηση, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να καλέσουμε τον Αντιπρόεδρο στην συζήτηση που θα έχουμε με ναι. τα Εθνικά Κοινοβούλια για την έκθεση προόδου. Δεν το συμπεριέλαβα, συμπεριέλαβα συγγνώμη, στην ερώτησή μου γιατί δεν είχα χρόνο, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση που θα γίνει για την έκθεση Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να είστε παρόν. Βεβαίως αν προτιμάτε μπορείτε να τα πείτε κατευθείαν με την Πρόεδρο, αλλά εμείς με μεγάλη χαρά θα σας υποδεχτούμε πάλι εδώ. Σε δύο λεπτά συνεχίζουμε. Dear, to Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με την ανταλλαγή απόψεων που αφορά την έκθεση του Σφεν Γκίγκολτ. Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε οργανώσει και μία ακρόαση από κοινού με την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, Ελέγχου του Προϋπολογισμού και θεωρώ ότι και για τον ΣΦΕΝ αλλά και για την έκθεση αυτή η ανταλλαγή απόψεων και ακρόση ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Ξεκινάμε λοιπόν και δίνω εκ νέου τον λόγο στον ΣΦΕΝ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την έκθεση. Δεν πρόκειται για συναισθήματα, όπως ε, ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Πρόκειται για γεγονότα, για το γεγονός ότι κάποιοι πολίτες τα τελευταία χρόνια έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και βλέπουμε πολλές χώρες, βλέπουμε πολιτικά κόμματα, κινήματα να χρησιμοποιούν αυτήν την νέα κατάσταση και να στηρίζουν διάφορους λόγους που βασίζονται στο λαϊκισμό και σε εσφαλμένα επιχειρήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι το θέμα της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ακαιρεότητας στους θεσμούς και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι επειδή τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χαμηλότερο επίπεδο διαφάνειας και ακαιρεότητας. Αντίθετα, έχουμε υψηλότερα. Αλλά το ε, αίσθημα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι βρίσκονται μακριά από την Ευρώπη και ότι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους μακριά, κάπου μακριά στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, δεν λογοδοτούν σε κανέναν. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι αυτή η λογοδοσία δεν υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη πραγματικά, και αυτό είναι απέτηση των δημοκρατικών πολιτευμάτων, να απαιτήσουμε υψηλά επίπεδα λογοδοσίας, διαφάνειας και ακεραιότητες. Μετά λοιπόν από συζητήσεις, ανταλλαγές απόψεων, workshops, ακροάσεων, επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλες διευθύνσεις, την Επιτροπή. Και φυσικά εδώ δεν θα σας παρουσιάσω όλες τις προτάσεις τις οποίες ε, διάβασα και προσπάθησα να ενσωματώσω. Αλλά είμαι πολύ περίεργος αν θέλετε και έτοιμος να ακούσω τις δικές σας προτάσεις. Ακούσατε τι είπε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τα λόμπι, για τις ομάδες συμφερόντων. Και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι όχι να συζητήσουμε για τα προσωπικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα των μεν και των δεν και όλων των εμπλεκόμενων στην ομοθετική διαδικασία. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε αυτοί οι οποίοι συναντούν οργανωμένες ομάδες συμφερόντων να γνωρίζουν σε ποιον μιλούν και να ενημερώνουν το κοινό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιους συναντάμε και ποια συμφέροντα εκπροσωπούν. τα αντικρουόμενα συμφέροντα είναι μια πραγματικότητα. Και οι διαδικασίες, αν θέλετε, δεν είναι ικανοποιητικές, γιατί αυτοί που αποφασίζουν για τα αντικρουόμενα συμφέροντα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι ίδιοι μέλη του Κοινοβουλίου. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων πολύ συγκεκριμένη. Πώς μπορεί κάποιος να αξιολογήσει και να εκφράσει άποψη για συναδέλφους που βρίσκονται στην ίδια πολιτική ομάδα με εσάς. Χρειάζονται εμπειρογνώμονες, εξωτερικοί, ανεξάρτητοι, ειδικοί για θέματα δεοντολογίας και αρχών. Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω αυτών των διαδικασιών που επαναλαμβάνω χωλένων. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο αυστηρούς κανόνες και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Αντιπρόεδρος δεν απάντησε στην ερώτησή μου όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για τους επιτρόπους. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι παραδείγματο χάρη στη Γενική Διεύθυνση για ε, τον ανταγωνισμό μπορεί κανείς να ασχοληθεί με μια υπόθεση συγχώνευσης και κατόπιν όταν πρόκειται για συγχωνεύσεις στον ιδιωτικό τομέα, καταλαβαίνετε ότι δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, οι οποίοι ισχύουν για δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές επιχειρήσεις. Μπορεί κάποιος παραδείγματο χάρη να ε, δουλεύει ταυτόχρονα και για μια ιδιωτική, έναν ιδιωτικό φορέα και να είναι μέλος εδώ μιας υπηρεσίας της Επιτροπής. Μπορεί μάλιστα να βρίσκεται και σε άδεια και ταυτόχρονα να συνεργάζεται με κάποιον ιδιωτικό ε, φορέα, ο οποίος εμπλέκεται σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να το επανεξετάσουμε. Η Ευρώπη ε, και εδώ θα αναφερθώ στην πρόσβαση στα έγγραφα, βρίσκεται την πρώτη γραμμή όσον αφορά τη διαφάνεια και την πρόσβαση. Έχουμε δικαίωμα, αν θέλετε, να ενημερωθούμε και έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλά όγραφα, τα οποία όμως πολλές φορές δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πούμε, δεν έχει τον κατάλογο των εγγράφων που έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρει, λοιπόν, κανείς πού να ψάξει και τι να βρει. Και όταν μιλάμε για διαδικασία νομοθετική και διαφάνεια, πιστεύω ότι μπορούμε σαφώς να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όλοι μας και κυρίως το Συμβούλιο. Πολλά συμβαίνουν στο Συμβούλιο τα οποία γίνονται χωρίς απολύτως καμία διαφάνεια. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί δικαιολογημένες ανησυχίες όταν παραδείγματος χάρη αναφερόμαστε στο ευρώ, στην ευρωζώνη. Όπως ξέρετε, το Eurogroup δεν έχει πρακτικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του αυτό. Και θα πρέπει να απαιτήσουμε από τους εταίρους μας να έχουν το ίδιο επίπεδο διαφάνειας όπως έχουμε και εμείς. Παραδείγματο χάρη για τους τριμερείς διαλόγους. Δεν νομίζω ότι πρέπει εδώ να μειώσουμε ή να περιορίσουμε την πρακτική των τριμερών διαλόγων. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιο ισχυρό σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία στην Ολομέλεια για να ενισχύσουμε και να ε, στηρίξουμε την ε, θέση μας. Αυτή όμως η τριμερή διάλογη είναι αδιαφανής. Χρειαζόμαστε λοιπόν και ένα μητρό για τους τριμερείς διαλόγους ενδεχομένως. Όταν συμβαίνουν συναντήσεις, ποιο συμμετέχει και τα πρακτικά θα πρέπει να δημοσιεύονται. Αυτό ακριβώς προτείνω. Όσον αφορά τώρα αυτούς που ενημερώνουν την κοινή γνώμη, τους whistleblowers, είναι πάρα πολύ σημαντικό ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προειδοποιήσεις που αφορούν τις χρηματαγορές θα πρέπει να τους προσφέρουμε προστασία και εκτός των συνόρων της χώρας τους. Θα πρέπει λοιπόν η οδηγία για αυτούς τους ανθρώπους που προειδοποιούν την κοινή γνώμη να ολοκληρωθεί και να στηριχτεί. Είδατε λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες στις προτάσεις και ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους σκιώδεις εισηγητές με τους οποίους έχω ήδη ανταλλαγές απόψεων οι γνωμοδοτήσεις των άλλων επιτροπών που έχουν ε, σαφώς ε, στηριχτεί στο μεγάλο ενδιαφέρον και βεβαίως πάρα πολλοί πολίτες. Εκατοντάδες ε, μου έστειλαν μέσω της ιστοσελίδας προτάσεις θα συνεχίσω λοιπόν να τις επεξεργάζομαι και με μεγάλη χαρά θα συνεχίσω την συζήτηση μαζί σας. Είναι σίγουρα οι προτάσεις μου, προτάσεις οι οποίες θα προκαλέσουν συζήτηση, αλλά θεωρώ ότι το θέμα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακαιρεότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους δεν ξέρω αν κάποιος αντικαταστάθηκε με κάποιον άλλο. Ας ε, μου το γνωστοποιήσει. Αρχίζουμε με το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Ντανούτα. Και ευχαριστώ πολύ το Σβέν, τον εισηγητή μας, για αυτό την ε, σημαντική έκθεση σχετικά με την διαφάνεια, την λογοδοσία και την ακαιρεότητα που προσφέρει μια μοναδική ε, ευκαιρία για καλή προσέγγιση για να βελτιώσουμε τα πρότυπα ε, και στους τρεις ε, τομείς είμαι ευγνώμων για την προπαρασκευαστική εργασία που έγινε προτού παρουσιάστε την εισήγηση για πρώτη φορά τυπικά στην Επιτροπή ΑΦΚΟ και νομίζω ότι τα εργαστήρια που είχαμε με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού αρμοδίων ευρωβουλευτών και αξιωματούχων των οργάνων ήταν μια χρήσιμη άσκηση ε, σχετικά με την εισήγηση αυτή. Εφόσον πολλοί πρωταγωνιστές συμμετέχουν στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων θα πρέπει η διαδικασία αυτή να είναι όσο διαφανέστερη γίνεται για να καταλάβουμε ε, καλά το νόημα της αρχής της διαφάνειας έτσι όπως αναφέρεται στις συνθήκες. Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι ουσιαστικές αρχές για να υπάρξει ε, οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους Εβραίους ε, πολίτες ούτως ώστε να έχουμε νομιμότητα. Οι ε, πολίτες θα πρέπει να έχουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας ε, και αυτή η εισήγηση είναι, έχει αυτή την πρόθεση ε, για την νομοθετική εργασία και την νομιμότητα σχετίζονται με την διαφάνεια, την λογοδοσία και την ακαιρεότητα. Γι' αυτό ε, το ΕΛΚ θα είναι ανοιχτό και θα δεσμευτεί για το θέμα αυτό. Είναι ουσιαστικό να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα στη διαφάνεια και άλλες ε, αρχές ε, και αξίες στην εργασία των θεσμών μας. Νομίζω ότι από ορισμένε απόψεις το σχέδιο εισήγησης πάει πολύ μακριά και υιοθετεί μια ευρύτατη εφαρμογή της αρχής λαμβάνοντας υπόψη άλλες ε, αξίες, ε, οι οποίες όμως θα μπορούσαν ε, να απειλούνται. Υπάρχουν και επίμαχα θέματα σχετικά με ορισμένες προτάσεις που περιλαμβάνονται τώρα στο σχέδιο εισήγησης. Δεν μας φαίνεται αποδεκτό η δυνατότητα των ψηφοφόρων να έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο χωρίς φόρτο γραφειοκρατικό. Ε, το θέμα των διαπραγματεύσεων, ε, το απόρριτο των διαπραγματεύσεων ε, με τρίτους, όπως οι τριμερείς διάλογοι που αναφέρθηκαν στις παρατηρήσεις του κυρίου Γκίγκολτ. Επίσης, η αρχή της διαφάνειας, αν γίνει πολύ ευρεία, θα πρέπει όμως να διαφυλάσει και την δικαίωμα ιδιωτικότητας των μελών οι υψηλοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να αναμειγνύονται στις δημοκρατικές ευθύνες των μελών. Το να μην μπορεί κανείς να συναντήσει κανέναν άλλον εκτός από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό και να καταγράφεται διαδικτυακά η συνάντηση, ίσως αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Αυτά είναι τα θέματα, ε, τα στοιχεία που θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να φτάσουμε σε λύση και συμβιβασμό. Το θέμα που αναφέρθηκε στην προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο Τίμερμαντς, ε, το θέμα της υποχρεωτικής μεταβατικής περίοδου cooling off για τους επιτρόπους, τους ευρωβουλευτές ε, και το προσωπικό δεν είναι τελείως αναλογική αυτή η πρόταση παρόλο που η ευθύνη αναγνωρίζεται για όλους ε, θα προσπαθήσουμε λόγους, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ισορροπία, ε, συμβιβασμό με διάλογο με τον εισηγητή και τους άλλους χειώδεις εισηγητές των άλλων ομάδων για να καταλήξουμε σε μια καλή λύση ανάμεσα στις δύο απόψεις που σκιαγράφησα είναι προφανές ότι είναι πράγματι σημαντικό ε, να αυξήσουμε το επίπεδο διαφάνεια στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η εργασία των οργάνων γίνεται με τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους εταίρους μας στον κόσμο και εδώ αναφέρομαι σε πολύ λεπτές διαπραγματεύσεις που έχουμε, εκ των οποίων η πιο σημαντική και, είναι, ε, η οποία θέτει ερωτήματα για τη διαφάνεια είναι η εταιρική σχέση TTIP και εδώ ως πρώην διπλωμάτης θα πρέπει να, να πω ότι αν όλα μεταδίδονται αμέσως ε, διαδικτυακά, ε, τώρα αυτό θα πρέπει να αποδείξει ότι έχετε κερδίσει τις διαπραγματεύσεις. Για να έχουμε σοβαρές διαπραγματεύσεις αλλά και κατάλληλη ενημέρωση και εν ευθέτω χρόνο, η ισορροπία αυτή ανάμεσα στα δύο είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά ε, χρόνια και όταν θα έχουμε τις ε, συζητήσεις θα πρέπει η ομάδα να έχει τον χρόνο να ενημερώσει όλους τους άλλους συναδέλφους που δεν είναι εδώ σήμερα. Ε, τον κάθε ευρωβουλευτή, την κάθε ομάδα ε, και όταν θα συζητήσουμε ο Σβέν και εγώ Ίσως θα μπορούσαμε να παρατείνουμε το χρόνο για την κατάθεση τροπολογιών μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου διότι έχουμε και τις διακοπές, δύο-τρεις εβδομάδες δεν θα με την προσοχή μας στο θέμα αυτό. Έτσι, αν έχουμε το τέλος Φεβρουαρίου θα μπορούμε να έχουμε καλές προτάσεις και τροπολογίες και είμαι ανοιχτός σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για να έχουμε ένα καλό κείμενο που θα είναι σημαντική συνεισφορά στην διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτού συνεχίσω με τους σκιώδεις να πω δύο πράγματα. Πρώτον, στους βοηθούς και συμβούλους συναδέλφων που δεν είναι εδώ, να ξέρουν ότι η συζήτηση Μπρέσομπρόκ θα γίνει αμέσως μετά από αυτή τη συζήτηση και όχι το απόγευμα. Και έχουμε 25 λεπτά για να κλείσουμε τη συζήτηση Έχουμε πάρα πολλούς σκιώδεις που θέλουν να μιλήσουν και άλλους ε, υποψηφίους σύντομα. Λάινεν θα μιλήσει σαν σκιώδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τον Σφεν για την εξαιρετική του εργασία και για την ε, ε, διοργάνωση των workshops, το συντονισμό των συζητήσεων είναι βασική αρχή, θεμελιώδη, θεμελιώδης αρχή, αν θέλετε, της εργασίας μας, αλλά και σημαντικός παράγοντας για την εμπιστοσύνη των πολιτών, η διαφάνεια, η ακαιρεότητα και η λογοδοσία. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποφύγουμε να υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και ημών. Βρισκόμαστε μακριά, οι Βρεξέλλες και η Ευρώπη φαίνεται να βρίσκονται μακριά, γι' αυτό και τα επίπεδα και οι προδιαγραφές που θέτουμε για να υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία και κυριότητα πρέπει να είναι υψηλότερα και αυστηρότερα όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Συμφωνώ λοιπόν με τα περισσότερα μέτρα. Θεωρώ ότι αυτό που απαιτούν πλέον οι περισσότεροι πολίτες διαφάνεια μέσω του διαδικτύου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ενισχύσουμε. Η απώλεια εμπιστοσύνης είναι κάτι που δυστυχώς παρατηρείται σε πολλά μέρη της Ευρώπης από πολλούς πολίτες. Η οικονομική κρίση με την απώλεια πολλών θέσεων απασχόλησης, η κρίση με τους πρόσφυγες, η παγκοσμιοποίηση. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες νιώθουν ότι η Ευρωπή πλέον δεν τους προστατεύει από όλα αυτά τα φαινόμενα. Αυτό είναι όμως μια μονομερής, αν θέλετε, ε, αντιμετώπιση. Την ίδια ώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ενίσχυση της δαφάνειας σίγουρα θα δώσει σε πολλούς Ευρωπαίους πολίτες το συνέστημα ότι η Ευρώπη κάνει κάτι, τους ενημερώνει ότι έχουν πρόσβαση και βεβαίως θα πρέπει κανείς να προχωρήσει συγκεκριμένα για να βελτιώσει αυτήν την κατάσταση εμπιστοσύνης και έλλειψη εμπιστοσύνης. Όσον αφορά τη διαφάνεια, μιλήσαμε και με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς. Βεβαίως, εδώ θέλουμε όσον αφορά το Μητρό, να ολοκληρωθεί, να καλυφθούν τα κενά, να γίνουν πιο αυστηροί και πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι. Είμαστε βεβαίως ε, επίσης πάρα πολύ ανήσυχοι όσον αφορά και την ποιότητα των δεδομένων, των πληροφοριών και των στοιχείων που βρίσκονται σε αυτά τα Μητρώα. Και πιστεύω ότι για όλα αυτά χρειάζεται μια ε, σοβαρή δημόσια συζήτηση. Μιλήσαμε λοιπόν ε, σε πολλά επίπεδα για την ε, διαφάνεια. Πιστεύω ότι και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του TTIP, αλλά και σε άλλες διεθνείς συμφωνίες, συμφωνίες που έχουμε για οικονομικά εμπορικά θέματα με τρίτες χώρες, δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά και κλεισμένων των θυρών και χωρίς κανείς να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Χρειάζεται διαφάνεια. Πρόκειται για κάτι που θα επηρεάσει πλευρά την ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Το θέμα τώρα των τριμερών διαλόγων. Βεβαίως στην πράξη χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια για αυτούς τους τριμερείς διαλόγους και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε κάθε φορά που υπάρχει τριμερής διάλογος να υπάρχουν πρακτικά και από μέρους του Συμβουλίου έτσι ώστε να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να παρακολουθούν τι γίνεται και στις Ευρωπαϊκές Συνόδους Κορυφής και στα Eurogroup όποτε συνεδριάζουν. Θεωρώ λοιπόν ότι και για το θέμα της διαφάνειας αλλά και για το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν ε, πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομίζω ότι εδώ Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε γιατί είναι ίσως λίγο παρακινδυνευμένο να ζητήσουμε ο Ευρωβουλευτής να μην έχει απολύτως καμία άλλη δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Κάπως θα πρέπει να το προσδιορίσουμε αυτό. Ο Σβέν Γκίγκολτ όταν αναφέρεται στην αυτονομία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Έχω την εντύπωση ότι κάνει κάποιες λίγο υποχωρητικές προτάσεις. Δεν μπορούμε εμείς από μόνοι μας να πάρουμε αποφάσεις που μας αφορούν. Ζητάει μια συμβουλευτική επιτροπή. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει ίσως να το συζητήσουμε περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να αποφασίσει για αυτά τα θέματα αυτόνομα και μόνο του. Τα ευρωπαϊκά κόμματα, χαίρομαι ότι υπάρχουν τόσο πολλά ευρωπαϊκά κόμματα, αλλά στην τελευταία αναθεώρηση βλέπω και διαβάζω πολύ συγκεκριμένα τις προτάσεις που βρίσκονται στο σχέδιο της έκθεσης να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή και όσον αφορά βεβαίως την κατανομή της ε, χρηματοδότησης, της υποστήριξης που δίνεται στα πολιτικά κόμματα. Βεβαίως αυτό νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να συζητηθεί. Αυτό είναι ένα θέμα που φυσικά ενδιαφέρει όλο το Κοινοβούλιο, όλους τους συναδέλφους. Καταλαβαίνετε ότι όλοι θα δουν τι κάνει η Επιτροπή μας όταν συγκεκριμένες προτάσεις μπορεί να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα υποστηρίξω την πρόταση του κυρίου Γκίγκολντ. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε κάποιες αξίες πολλές φορές διαφορετικές μεταξύ τους. Στην στην φάση του τριμερούς διαλόγου ακούστηκαν διαφορετικές θα έλεγα αντιλήψεις για τη διαφάνεια εις βάρος ίσως μερικές φορές της ποιότητας της ε, νομοθεσίας. Νομίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος να φανούμε ιδιαίτερως υπερβολικά θα έλεγα πατερναλιστές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας χαρακτηρίζει και στις σχέσεις μας με τα εθνικά κοινοβούλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι απαραίτητη η συζήτηση την οποία κάνουμε στην παρούσα φάση. Νομίζω ότι μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την ποιότητα, την ειλικρίνεια των ηγετών μας των πολιτικών, την ποιότητα των πολιτικών μας θεσμών και λειτουργιών. Ένα από τα βασικά θέματα της έκθεσης αυτής είναι ότι δεν έχει ταμπού. Θέτει όλες τις ευαίσθητες ερωτήσεις και αυτό έχει μεγάλη μα πολύ μεγάλη σημασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο να είναι λειτουργικό και απαιτητικό. Έχουμε τα στοιχεία, βρισκόμαστε όλοι εδώ τώρα για να τα συζητήσουμε και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να μην μείνουμε στα λόγια και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πραγματικά αυτά τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον εισηγητή έτσι ώστε και οι υπόλοιπε κοινοβουλευτικές επιτροπές να προσφέρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Σόλτς. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση αυτή που μας έκανε, πώς ξεκίνησε, γιατί είναι σημαντική αυτή η έκθεση και βεβαίως έχουμε ξεκινήσει μεταξύ σκιωδών ε, ανταλλαγή απόψεων εδώ και πολύ καιρό, γιατί βεβαίως θα συνεχιστεί. Θα αναφερθώ σε τρία μονοσημεία, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω. Στην έκθεση αυτή μιλάμε βεβαίως ε, και για την έλλειψη εμπιστοσύνη, αλλά και για την καθοδήγηση και την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δηλαδή, βλέπετε ότι σήμερα υπάρχει πληθώρα νομοθετικών κειμένων και δεν υπάρχει πολιτική κατεύθυνση, δεν ξέρουμε πού πάμε. Ε, αν εκεί προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε σε περισσότερη διαφάνεια, για μένα έχουμε πετύχει πάρα πολύ ε, μεγάλα βήματα. Διαφάνεια λοιπόν, αλλά διαφάνεια επί της ουσίας. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι καθοριστικό για να επανέλθει η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Πώς ε, ε, επίσης θα μπορέσουμε αυτά τα μητρώα να τα κάνουμε δεσμευτικά. Δεν ξέρω, άκουσα κάποιες προτάσεις, ε, άκουσα και αυτά που προτείνει ο Σβέν, αλλά και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί παραπάνω. Τρίτο σημείο, οι διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα θεωρήσεων, θέματα που αφορούν άλλες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέματα ανάπτυξης, παραδείγματος, αναπτυξιακή πολιτική. Και η εντολή διαπραγμάτευσης για όλους αυτούς τους τομείς. Νομίζω ότι η απάντηση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής εδώ ε, δεν ήταν ε, σαφής. Καθότι Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Επιτροπή, όμως τα θέματα αυτά τα χειρίζεται το Συμβούλιο. Οι εντολές αυτές δίνονται από το Συμβούλιο για αυτό το είδος οι διαπραγματεύσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εδώ να στυλώσουν τα πόδια και να πούν ότι χρειάζεται μεταστροφή. Αυτή η πρακτική δεν μπορεί να συνεχιστεί. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα γιατί ξέρω ότι για όλα αυτά τα σημεία και για πολλά άλλα θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τον εισηγητή. Thank you. Understand that Ευχαριστώ. Ναι, ο Χαβιο Καστάντο δεν είναι εδώ. Κανείς δεν ε, είναι εδώ. Περνάμε στην Μπάρμπαρα. Ε, Μπάρμπαρα. Δεν ακούει η Μπάρμπαρα. Θέλεις να λάβεις τον λόγο Μπάρμπαρα. Όχι. George. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συγχαίρω τον κύριο Γκίγκελντ που συνέταξε ε, μια πολύ σημαντική εισήγηση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος διότι βλέπω ότι περνάει ο χρόνος. Πρώτα απ' όλα, αν τον κατάλαβα καλά, υποθέτει ότι όσο ψηλότερη είναι η διαφάνεια, τόσο ψηλότερη θα είναι και η εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τελείω σωστό. Υπάρχει ένα συσχετισμό, αλλά υπάρχουν και άλλε περιστάσει, άλλοι παράγοντε που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και που έχουν να κάνουν επίση με την, την αρχή ε, και, και επίσης με αποτελέσματα, την επιτυχία. Και τρίτον, ποτέ μην υποτιμάτε το γεγονός της κινησμού, δηλαδή την στάση πολλών που μπορούν ποια, αν όλα αυτά δημοσιοποιούνται, ποια είναι η πραγματική ιστορία πίσω από αυτά. Και υπάρχει μια σύγχυση στη σχέση ανάμεσα στην ε, εμπιστοσύνη και στη διαφάνεια. Ο κύριος Γκίγκολτ μίλησε για την διαφάνεια, λογοδοσία και κεραιότητα Και εγώ ε, θα προσέθετα και το feedback, ε, δηλαδή η διαδικασία πολιτικής για την οποία μιλούμε μπορεί να βελτιωθεί με ε, συνεισφορές από πάρα πολλές πηγές, ε, ποικίλε πηγές. Αυτό είναι το τρίτο μου σημείο. Εδώ υπάρχει μια ανάμεσα στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων, των διαφερομένων ε, και την ανάρμοστη επιρροή ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό το κίνδυνο. Μερικοί των λόμπι είναι πάρα πολύ καλοί και προωθούν τα συμφέροντά τους και ίσως οι συνομιλητές τους δεν είναι τόσο επιτυχημένοι όσο θα μπορούσαν να είναι. Σχετικά με το cooling off, τη μεταβατική περίοδο, έχω μια ερώτηση που είναι αρκετά δύσκολη. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Σβεν ότι δηλαδή ε, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στα δημόσια λειτουργήματα δεν πρέπει να μεταφέρονται στο ιδιωτικό τομέα. Τι γίνεται με αυτές τις γνώσεις, χάνονται ίσως αυτές οι γνώσεις. Ε, μια απώλεια υπάρχει. Αν κάποιος παραδείγματος χάρη ε, έχει αποκτήσει γνώσεις σε όργανα των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μεταφέρει τις γνώσεις αυτές στη χώρα του και να τις χρησιμοποιήσει εκεί. Αυτό είναι δύσκολο ερώτημα και ένα τελικό σημείο για τους whistleblowers, τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι παίζουν ε, ρόλο αλλά ε, μπορούν επίσης όμως να είναι επιφανειακοί, ανόητοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Μας προτείνει ένα κείμενο πλήρες, ισχυρό. Ο δικός μου σκιώδης εισηγητής ασχολήθηκε με τα πιο καθοριστικά από τα θέματα. Επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα να κάνω μόνο μερικές παρατηρήσεις σύντομα. Η πρώτη, έχει σχέση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ιδέα μιας συμβουλευτικής επιτροπής με πλειοψηφία μελών εκτός, εξωτερικών μελών. Και μείωση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου σε σχέση με την ε, υιοθέτηση των τελικών αποφάσεων για τον κώδικα συμπεριφοράς. Πάνω σε αυτό έχω πολλές αμφιβολίες. Θεωρώ ότι μία από τις βασικές αρχές των δημοκρατικών συστημάτων είναι το δικαίωμα αυτοδιοργάνωσης των κοινοβουλίων και του ελέγχου επίσης του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν. Η διαφάνεια είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν υπάρχουν λάθη θα πρέπει να είναι προφανή τα λάθη αυτά τα οποία, ε, για τα οποία θα μας ελέγξουν οι συμπολίτε μας και το να μεταφέρουμε αλλού αρμοδιότητες χαρακτηριστικές των κοινοβουλίων θα έλεγα είναι κάτι που με ενοχλεί. Το θέμα τώρα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Το να υπάρξει ένα έλεγχο της ορθότητας των προϋπολογισμών από μια ελεγκτική αρχή ανεξάρτητη αυτό είναι σαφές. Από την άλλη πάλι το κοινοβούλιο είναι συναρμόδιο για τον προϋπολογισμό και δεν μπορεί να μεταφέρει και να δώσει αλλού τις αρμοδιότητες του αυτές. Όσο περισσότερο αυξάνουμε την ε, δυσπιστία απέναντι ημών των ιδίων, το ίδιο κάνουν και οι πολίτες και όχι το αντίθετο. Υπέρ της διαφάνειας μεν, κατά της δυσπιστίας δε. Αυτό ισχύει για όλους, ισχύει γενικότερα, δεν είναι ένα θέμα μιας πολιτικής ή μικροπολιτικής για το Κοινοβούλιο. Κυρία Γκουλάρ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάνει εξαιρετική δουλειά ο εισηγητής. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να πιέσουμε λίγο περισσότερο εδώ. Έρχομαι πάνω σε αυτό το οποίο είπε η Μεσέδες. Είχαμε πάει με τον Πασκάλ Τυρό σε μια ραδιοφωνική εκπομπή προηγουμένως. Δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την συστηματική δυσπιστία εις βάρος του Κοινοβουλίου. Έχω βαρεθεί την αυτομαστίγωση. Λες και στις εθνικές ε, οργανώσεις, της χώρες μας υπάρχουν μόνο κάποιοι Άγιοι οι οποίοι ούτε λόμπι υφίστανται, ούτε επηρεάζονται. Λοιπόν, Σίγουρα έχουμε να κάνουμε με ένα στοιχείο το οποίο από το τοπικό επίπεδο μέχρι το ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλα τα επίπεδα δημόσιας οργάνωσης απαιτείται να υπάρχει διαφάνεια. Πόσο μάλλον που εγώ δεν νομίζω και είμαι ειλικρινής εδώ αλλά και κοινική δεν νομίζω ότι υπάρχουν επακριβή συστήματα. Ο Λόρδος Χιλ το είπε στην ακρόαση που οργάνωσε και το είδα εγώ παίρνοντα το θαλής. Ο Λόρδος Χιλ είπε «Μπορούμε να υποχρεώσουμε τους βουλευτές ε, να έχουν ένα κατάλογο των ανθρώπων ε, που συναντούν στο γραφείο τους. Αλλά όταν βλέπετε κάποιους και συναντάτε και μιλάτε με κάποιους στους διαδρόμους του τρένου ας πούμε, τι κάνετε. Λοιπόν, μην έχουμε την ψευδέστηση ότι εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κλειστό τέλειο σύστημα και να μην θεωρήσουμε ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πιο καθαρό, είναι πιο clean από ό,τι τα υπόλοιπα επίπεδα λήψεως αποφάσεων. Τώρα, ε, για κάποια σημεία που έθεσε ο κύριος Σόλτς. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο. Υπάρχει το θέμα των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων, όχι μόνο εμπορικών διαπραγματεύσεων θα έλεγα, αλλά γενικά των διεθνών διαπραγματεύσεων. Τι θέλουμε εμείς να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο τι γίνεται. Άκουσα ότι στο TTIP στην αρχή υπόθηκε σε ορισμένες χώρες ότι θα συμμετέχουν και βουλευτές. Τότε που είναι ο διαχωρισμός των εξουσιών. Η διπλωματία έχει μια τάση να λειτουργεί κρυφίως σε ορισμένες περιπτώσεις. Σωστά ή λάθος. Είναι σωστό να πούμε ε, ότι υπάρχει υπερβολή σε επίπεδο διακυβερνητικό ε, και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις 19 χώρες από τη μία και στις 28 από την άλλη. Αλλά δεν πρέπει να γενικεύουμε. Αυτά τα οποία συμβαίνουν ας πούμε σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών συζητώντας θέματα όπως η Τουρκία σαν παράδειγμα, κανένα δεν ξέρει τίποτα. Λοιπόν, μια πρώτη παρατήρηση που ίσως ακουστεί κάπως ε, προκλητική. Τρία χρόνια κούλιμοφ. Τρεις ολόκληρες χρονιές είναι υπερβολικό. Θα πρέπει ε, να προσπαθήσουμε να δούμε τι γίνεται στη σχέση δημόσιος και ιδιωτικός τομέας και να μην αποκλειστούμε από το, ε, από το περιβάλλον μας. Για σκεφτείτε όλους ε, όσους τους νέους που παίρνουν μία σύμβαση τριετίας Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να αλλάξει, θα είναι άδικο απέναντι στους νέους. Προφανώς θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για τους επιτρόπους και λιγότερο δεσμευτικές ρυθμίσεις για αυτούς που είναι σε χαμηλότερο επίπεδο. Πρώτον, θα ήθελα επίσης να δούμε και σε ποιο βαθμό ήταν αρνητική μέχρι τώρα η επικουρικότητα. Ο Σβέν θα το αγαπήσει αυτό. Όταν δούμε σαν παράδειγμα τα προβλήματα διαφθοράς ε, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ταμεία, αυτό γίνεται και σε επίπεδο δημοτικών και εθνικών αρχών. Λοιπόν, η, η διαχείριση του προϋπολογισμού στην ουσία εκχωρείται σε διοικητικές δομές πάνω στις οποίες έχουμε ελάχιστο έλεγχο. Αυτό πρέπει να το πούμε όταν βλέπουμε ότι στην Πολωνία έχουμε πλέον μια κυβέρνηση η οποία παίρνει το 4% του ΑΕΠ της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφαιρεί ε, τις σημαίες ε, πίσω από τις ομιλίες της Πρωθυπουργού. Λοιπόν, τίθεται θέμα ακαιρεότητας, τίθεται θέμα ειλικρινίας, τίθεται θέμα ε, για τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες. Είμαστε πρότυπο διαφάνειας εγώ είμαι υπέρ της χρήσης του συστήματος δεχόντι για την κατανομή των θέσεων. Ξέρω ότι έχουν γίνει ολόκληρες ιστορίες για τους λεγόμενους σπίτσεν, τα κτλ. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο διανέμουμε ε, τις ε, θέσεις ανάλογα με την εθνικότητα, αυτό τώρα είναι σωστό, είναι διαφανές, είναι ακέραιο. Δεν μπορούμε εμείς να δίνουμε μαθήματα σε κανέναν και ταυτόχρονα να μην προσπαθούμε να καταστήσουμε διαφανή τις σχέσεις μας στο εσωτερικό της διάσκεψης των Προέδρων, ε, όταν κατανέμονται οι αρμοδιότητες ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ιεραρχία η πολιτική σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Πρέπει να γίνει μια γενικότερη συζήτηση γύρω από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ρίτσαρτ. Ευχαριστώ, συγχαίρω τον εισήγητη που μας έβαλε τόσα πολλά επιτάπητος για να τα εξετάσουμε τέσσερα σημεία σχετικά με τα σχόλιά σας σχετικά με τις συμφωνίες πρώτης ανάγνωσης τα εξετάζουμε επίσης και στην ομάδα εργασίας αυτής της Επιτροπής και συμφωνώ με την προσέγγισή σας ότι δεν είναι θέμα να απαγορεύσουμε συμφωνίες πρώτης ανάγνωσης αλλά θα πρέπει να γίνουν πιο διαφανείς και με ορισμένες βαλβίδες ασφαλείας. Ε, θα ήθελα να είμαι σύντομος, γι' αυτό δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δεύτερον, σχετικά με το θέμα του αν υπάρχει σύγκρουση συμφορώντων ε, ανάμεσα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς το αξιολογούμε αυτό. Είναι ενδιαφέρον το σημείο και θα ζητήσω από τον εισηγητή να δει τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε ανεξάρτητη αρχή η ανεξάρτητη αρχή ε, κοινοβουλευτικών προτύπων, όπου δεν είναι μέλη κοινοβουλίου που αξιολογούν μέλη κοινοβουλίου, αλλά εξωτερικοί παράγοντες. Ξέρω ότι ε, θα, δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μοντέλο για κάτι, αλλά θα πρέπει να το πω αυτό. Είναι κάτι το οποίο εισήφθηκε από την κυβέρνηση των εργατικών. Δεν είναι πρόσφατη αυτή η μεταρρύθμιση. Και αυτό είναι, αν θέλετε, μια απόδειξη ποιότητας. Τρίτον, το θέμα των ευρωβουλευτών που έχουν και άλλα επαγγέλματα, άλλες δουλειές. Είναι πολύ δύσκολη, παραμπτός χάρη για έναν αγρότη, να εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να πουλήσει το αγρόκτημά του. Ε, θα πρέπει να δούμε τη διατύπωση πολύ καλύτερα. Θα πρέπει να δούμε ε, τα μέλη που ενώ έχουν, είναι ευρωβουλευτές είναι σε μια εταιρεία που κάνει λόμπι, που ασκεί πίεση στο κοινοβούλιο. Ναι, ο κύριος Μπροκ πήρε το τηλέφωνο. Ε, το θέμα που των ευρωβουλευτών που δουλεύουν για ομάδες συμφερόντων ε, και που χρησιμοποιούν για κέρδος ε, τα στοιχεία, τις πληροφορίες τους και τις γνώσεις τους. Και θα πρέπει επίσης να ε, έχουμε επίσης τους κανόνες για δήλωση ενός, ενός συμφέροντος που υπάρχει πριν. Και εδώ ένας αγρότης θα πρέπει να πει ότι έχει συμφέρον να ψηφίσει γι' αυτό, διότι αυτό θα βοηθήσει την αγροτική μου επιχείρηση. Και ένα τελικό σημείο, τελευταίο σημείο, σχετικά με το αποτύπωμα. Πολλοί από εμά το κάνουμε αυτό, είναι πολύ εύκολο. Ε, μπορούμε να κάνουμε έναν κατάλογο των ποιον συναντούμε και να το βάλουμε ε, στο διαδίκτυο. Ε, βεβαίως λέει κανείς ότι η άσκηση είναι πάρα πολύ γραφειοκρατική, αλλά δεν είναι κάτι δύσκολο να γίνει. Και αυτό που είπε ο Φραν Τίμα μας προηγουμένως, μέχρι πού ε, θα προχωρήσει κανείς στην ιεραρχία στην Επιτροπή μέχρι ε, τα κατώτερα επίπεδα στελεχών. Αν υπάρχουν ανησυχίε για λόμπι, τότε πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Ε, αν κάποιος βγάζει κάποιον για γεύμα, ε, θα πρέπει αυτό να εγγραφεί, να καταχωριστεί. Δεν είναι θέμα για το πού βρίσκεται το, ο υπάλληλο στην ιεραρχία. Το θέμα είναι αν έχει υποστεί πιέσει από ομάδα συμφερόντων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τις προτάσεις του εισηγητή. Η εισήγηση ε, έχει κάποιες προτάσεις που θα μας επιτρέψουν να προοδεύσουμε στο θέμα της διαφάνειας μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εφόσον δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να προσθέσω ότι η συζήτησή μας πρέπει να μας επιτρέψει να διακρίνουμε τις καλές προτάσεις που θα μας επιτρέψουν να προωθήσουμε την διαφάνεια από τις πιο ριζοσπαστικές λύσεις και ίσως υπερβολικές που αυτές θα ενισχύσουν τη γραφειοκρατία, τις υποψίες, τις υπόνοιες ε, για τη θητεία μας χωρίς να επιλύουν πρακτικά τα προβλήματα. Οφείλουμε λοιπόν να βρούμε λύσεις ισορροπημένες. Να έχουμε ένα μητρό των ομάδων συμφερόντων είναι μια καλή ιδέα, αλλά να εμποδίσουμε ε, τον εισηγητή, τους εισηγητές να συναντούν με αυτούς που επιθυμούν να συναντήσουν επειδή ανήκουν σε ένα λόμπι, να ζητούν μηνιαίες εκθέσεις από τα λόμπι, να ζητούν από όλους τους επικέπτες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμπληρώνουν ένα έντυπο λέγοντας ότι ανήκουν σε ένα λόμπι, ίσως αυτό είναι υπερβολικό. Να ενισχύσουμε λοιπόν τους κανόνες για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην άσκηση του λειτουργήματος, είναι καλό να έχουμε λύσεις όπως η μείωση των όσων κάνουν ε, οι βουλευτές. Αυτό ίσως σε ένα χρονικό διάστημα, ίσως αυτό είναι υπερβολικό. Η διαφάνεια στην αποκάλυψη των εγγράφων, δημοσιοποίηση εγγράφων και πρακτικών είναι καλή ιδέα, αλλά το να πούμε ότι οι προπαρασκευαστικές συναντήσεις του Συμβουλίου θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, αυτό ίσως είναι υπερβολικό. Θα πρέπει λοιπόν στη συζήτηση αυτή να αναζητήσουμε ε, μια ισορροπία. Γι' αυτό και εγώ θα παρουσιάσω ε, τροπολογίες. Πασκάλ ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες εφόσον έχω πλήρη εμπιστοσύνη στον Σβέν για να υποστηρίξει την εισήγησή του. Θα ήθελα απλώς να απαντήσω στη Σιλβή και στη Μερσέντε για ένα θέμα αρχής. Ακούω ότι δεν θα πρέπει να ζητούμε περισσότερα από ε, το όργανο το ευρωπαϊκό από ό,τι θα ζητούσαμε από ένα κράτος. Αυτό ε, θεωρητικά είναι σωστό, αλλά στην πράξη δεν μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη τα θεσμικά όργανα τα ευρωπαϊκά είναι ε, το σημείο εισόδου των ιδιωτικών συμφερόντων, δηλαδή των λόμπι. Λυπούμε, λυπούμε πολύ, αλλά πρέπει να είμαστε παραδειγματικοί για τα θέματα αυτά, διότι στα εθνικά κράτη υπάρχει μια εικόνα ε, των πολιτών ότι υποστηρίζουν το δημόσιο συμφέρον. Εμείς έχουμε μια δυσκολία. Κανείς στην Ευρώπη δεν πιστεύει ότι τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα προστατεύουν το κοινό συμφέρον και το κοινό καλό. Λυπούμε, λυπούμε, ξέρω ότι δεν σας πείθω, αλλά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οφείλουμε ως Ευρώπη να δώσουμε το παράδειγμα για ορισμένα θέματα και το θέμα της ισορροπίας ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον, στο κοινό καλό και τα ιδιωτικά συμφέροντα είναι ένα θέμα σημαντικό. Η εμπειρογνωμοσύνη ανεξάρτητη είναι σημαντική. Αυτά είναι προβληματικά. Αν δεν τα αντιμετωπίσουμε στεναρά, άλλη μια φορά θα δούμε την ευρωπαϊκή ιδέα να οπισθοδρομεί δεν θα πρέπει να κάνουμε λάθος ε, νομίζοντας ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ομοθετούμε για το θέμα αυτό. Στρέν. Δύο λεπτά. μισή λεπτό. Βεβαίως δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε όλη τη συζήτηση τώρα. Θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα αυτό. Ίσως πρέπει να σταματήσετε να μιλάτε ή δεν ακούω τι λέω. Εγώ έχω χρόνο. Ίσως ο Έλμαρ Μπρόκ δεν έχει χρόνο. Δεν μπορώ βεβαίως να σχολιάσω όλα αυτά, για όλα αυτά που άκουσα, αλλά επί της ουσίας θα θέλω να πω το εξής. Κάποιες φορές βλέπω να έχουμε έναν περίεργο ιδεαλισμό όσον αφορά τη σχέση κράτους και πολιτών. Αυτό που λέτε είναι ότι τι ωραία που ήταν τότε που οι πολίτες μας πίστευαν, πίστευαν τις κρατικές αρχές και δεν χρειαζόμασταν διαφάνεια γιατί σήμερα που υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τη διαφάνεια και τα λοιπά και τα λοιπά, κατά κάποιο τρόπο κατατροπώνουμε αυτήν την ιδεαλιστική προσέγγιση ότι το κράτος προστατεύει ε, τα συμφέροντα των πολιτών και ότι έχει έναν πολύ ε, ιδανικό ρόλο. Σήμερα η εμπιστοσύνη υπάρχει, η δυσπιστία υπάρχει, η καχυποψία υπάρχει. Δεν χρειάζεται εμεί να τη δημιουργήσουμε. Υπάρχει. Είναι πραγματική και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι σημαντικό πριν πάμε στις λεπτομέρειες. Και αυτό ισχύει για όλα τα επίπεδα και για τις ομάδες συμφερόντων, τα λόμπι. Δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε εμείς καχυποψία επειδή θα αυξήσουμε την στήριξη, αν θέλετε, ε, και θα δημιουργήσουμε αυστηρούς κανόνες. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε ισορροπημένες προτάσεις και θα μπούμε στην συζήτηση όλων αυτών σημείο προς σημείο, αλλά ως προς την γενικότερη προσέγγιση πρέπει να είμαστε σοβαροί. Τώρα, για τα χρονοδιαγράμματα. Οι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες είπαν μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Άκουσα 19 Φεβρουαρίου από τη Γραμματεία για την προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Τέλος Φεβρουαρίου λέει το ΕΛΚ. Γιατί όχι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ και αν συμφωνείτε όλοι εγώ δεν είμαι κατά. Βεβαίως θα ήθελα να επανέλθουμε προς συζήτηση με το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή και βεβαίως όσον αφορά τις ε, τροπολογίες θα συνεχίσουν οι συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Θέλω να συζητήσω και με την αρμόδια ομάδα για να αποφύγουμε επικαλύψεις. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα σχόλιά σας και δέχομαι την πρότασή σας για αλλαγή της ημερομηνία για την υποβολή των τροπολογιών τέλος Φεβρουαρίου, εγώ δεν είμαι κατά αλλά θεωρώ επίσης ότι όλοι οι εκπρόσωποι πολιτών, φορέων που αφορούν ομάδες συμφερόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε εποφές μαζί τους. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν σήμερα, αν θέλετε, προτάσεις για να αποκλειστούν κάποιοι από το μητρέο των ε, ομάδων συμφερόντων, των λόμπι, να συνεχίσουν όμως να έχουν επαφές με τους ε, θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Σήμερα μπορώ να σας προτείνω μια νέα ημερομηνία για την υποβολή των τροπολογιών 29, 29 Φεβρουαρίου. 29 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Συμφωνείτε για τις τροπολογίες. 29 Φεβρουαρίου υπάρχει ως ημέρα. Υπάρχει. Το έχω ελέγξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Mercedes Μπρέσο Έλμαρ Μπρόκ. Θέλω επίσης να σας πω ότι θα διακόψουμε ακριβώς στις 12 και θα ψηφίσουμε στις 12. Γιατί αλλιώς θα μου πείτε ότι αλλάζουμε το πρόγραμμα. Έλμαρ ή η Mercedes. Ε, grazie, grazie Presidente. Ε, purtroppo... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και το κείμενο εργασίας μας περιλαμβάνει πάρα πολλά θέματα. Πάντως, να σας θυμίσω ότι τον τελευταίο καιρό υπήρξαν διαδοχικά ορισμένα γεγονότα ε, πρώτα η κρίση μεταναστευτική προσφυγική, μετά οι δραματικές επιθέσεις στο Παρίσι και αλλού. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάποιες από τις, ε, κάποια από τα στοιχεία της έκθεσης αυτής έχουν μεγάλη σημασία. Και δεν θα πρέπει να αναφερθούμε μόνο σε πιθανές αλλαγές των συνθήκων, αλλά να δούμε ακριβώς και τι δυνατότητες έχει η συνθήκη της Λισαβόνας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για μεγαλύτερη συνεργασία και αποτελεσματικότητα της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θέματα τα οποία μας αποσχόλησαν μέχρι τώρα ήταν θέματα πολιτικά κοινωνικά, ε, μετανάστες κτλ, ενώ τώρα μιλάμε κυρίως για θέματα ασφάλειας. Στόχος της έκθεσης αυτής είναι να δείξουμε με ποιο τρόπο η συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνει ένα τεράστιο δυναμικό που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να προχωρά στην ολοκλήρωσή της, εφόσον το επιθυμεί βέβαια, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις χωρίς να τεθεί άμεσα το περίπλοκο θέμα και ο χρόνος που απαιτείται για μία τροποποίηση των συνθήκων. Τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολλά. Δεν έχω τον χρόνο να ε, έλθω στην ουσία των προβλημάτων αυτών, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στα πιο σημαντικά. Καταρχάς η οικονομική διάσταση, την οποία δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ευάφηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες προφανώς στην παρούσα φάση είναι ανεπαρκής για να υπάρξει πλήρης ολοκλήρωση της Ένωσης και γι' αυτό προτείνουμε μια ολόκληρη σειρά από θέματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε και να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των πολιτών μας έτσι ώστε η Ευρώπη να επανέλθει στην ανάπτυξη στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη διασφάλιση της λειτουργίας των αγορών. Εντός του πλαισίου αυτού λοιπόν θα επιθυμούσαμε να υπάρξει ένα πραγματικό κοινωνικό σύμφωνο με προκαθαρισμένους δείκτες ισχυρούς και δεσμευτικούς, όπως ισχύει για τα δημοσιονομικά και τον προϋπολογισμό. Ένα άλλο θέμα είναι οι προκλήσεις οι στρατηγικές της εποχής μας, η ανάγκη κυρίως ανάπτυξης μιας κοινή εξωτερικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και όπως το δείχνει και το πρόσφατο αίτημα του Προέδρου Ολόντα για την ενεργοποίηση του άρθρου 42,7 των συνθήκων, υπάρχει χώρος παρέμβασης Υπάρχει και το 122 της Συνθήκης Λειτουργίας, το οποίο ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μια διαδικασία κοινή καταπολέμησης των τρομοκρατικών ενεργειών. Κάνουμε μια σειρά από προτάσεις λοιπόν, οι οποίες είναι θα έλεγα ισχύρες και ε, χρησιμοποιούνται εντός των συνθήκων. πέρα από το θεσμικό κομμάτι, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε συνδέεται και με τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου, που είναι το λιγότερο γνωστό και λιγότερο διαφανές όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέσαμε το θέμα αυτό ως προς την διαφάνεια. Για να το καταστήσουμε πιο διαφανές θα πρέπει επί μιας εθελοντικής βάσης να ε, μπορέσει να λειτουργήσει σαν, ένα πραγματικό, ε, σαν μια πραγματική γερουσία αν θέλετε ή άνω έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει και την δυνατότητα την οποία εμείς παρέχουμε σε επίπεδο προπαρασκευαστικό, προπαρασκευαστικών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει την διαφάνεια και την νομοθετική ευκρίνεια του τρόπου ε, λειτουργίας του Συμβουλίου. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόταση και τα οποία θα προσθέσει ο Μπροκ. Στη συνάντηση την οποία είχαμε την προηγούμενη φορά με τα κοινοβούλια των κρατών μελών μας υπογραμμίστηκε η ανάγκη η οποία υπάρχει να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εμπλέξουμε με καλύτερο αποτέλεσμα στην όχι άμεση νομοθετική διαδικασία αλλά στο, στην πορεία διαμόρφωσης των νομοθετικών προτάσεων πώς μπορούν να εμπλακούν καλύτερα τα κοινοβούλια των κρατών μελών και Γι' αυτό και τα κοινοβούλια θεωρούν με θετικό τρόπο ε, τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό όχι μόνο σε αρνητικό επίπεδο με τις κίτρινες και κόκκινες κάρτες αλλά θετικά και επικοδομητικά. Πρέπει να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτή την θέλετε ερώτηση. Παραμένει λοιπόν και τελειώνω το πρόβλημα εμπόδιο μεγάλο που είναι η ψήφος με ομοφωνία, είναι μια τροχοπέδη στην ε, νομοθετική διαδικασία, είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί όλο και περισσότερο σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση αμυγός διακυβερνητικού χαρακτήρα. Η βασική ανησυχία η οποία βρίσκεται στη βάση της έκθεσής μας είναι να επιστρέψουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να βασίζεται στην κοινοτική μέθοδο και όχι να επιλέγουμε κάθε φορά διακυβερνητικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Ο Έλμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. πολύ σύντομα Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, δεν θα επαναλάβω όλα αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο έγγραφο εργασία. Γνωρίζουμε όλοι τι πρωτοβουλίε μα. Η πρότασή μα είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτά που προέρχονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια θα προέρχονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια και βεβαίω ε, εμεί ε, θα κάνουμε τι δικέ μα. Ε, θα συνεχίσουμε να έχουμε τι δικέ μα αρμοδιότητε. Τι επόμενε ημέρε βεβαίω θα προετοιμάσουμε το τελικό σχέδιο και ελπίζω μέχρι την μεθεπόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο να είναι έτοιμο έτσι ώστε αρχές Ιανουαρίου να μπορέσει να γίνει η παρουσίαση της, ε, του σχεδίου έκθεσης και να μπορέσουμε να τηρήσουμε και την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Άλλη μια εβδομάδα λοιπόν είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και βάσει αυτών που θα λάβουμε θα προετοιμάσουμε με τη γραμματεία το κείμενο, το τελικό ε, κείμενο σχέδιο. Είναι πολύ συγκεκριμένος, αν θέλετε, ο σκοπός μας να παραμείνουμε στα πλαίσια της συνθήκης. Σας παρακαλώ, οι υπόλοιπες προτάσεις να σταλούν στον κύριο Φερχόφστα, το έχει σε εμάς. Θα περιοριστούμε με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο στο εσωτερικό της συνθήκης. Αυτά δηλαδή που μπορεί να υλοποιηθούν, που μπορεί να πραγματοποιηθούν. Εντάξει, σας παρακαλώ πολύ, μην προσπαθείτε να ε, παρεκκλίνετε και να ξεπεράσετε τα όρια των συνθήκων. Βέβαια, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να συζητηθούν, γιατί έτσι και όχι αλλιώ. αλλά ε, εμείς ε, θέλουμε να είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το όριο αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Ναι, και εμείς και η Επιτροπή. Δεν μπορούμε ε, εδώ να επεκτείνουμε παραπάνω τα θεσμικά μας όρια και βεβαίως αυτά σε σχέση με την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της επικουρικότητας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, αυτές οι δύο αρχές ισχύουν και εμείς τις στηρούμε. Ευχαριστώ πολύ πραγματικά για όλες τις προτάσεις ε, που λάβαμε και που ενδεχομένως θα λάβουμε ακόμα. Υπάρχουν ε, σίγουρα παραδείγματο χάνει για την πορτοκαλί κάρτα διάφορα θέματα που θα συζητηθούν ε, και στα πλαίσια του δημοψηφίσματος που θα λάβει η χώρα στη Μεγάλη Βρετανία για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ε, υπάρχουν πολλά θέματα που συμπεριλαμβάνονται ή δεν συμπεριλαμβάνονται. Το άρθρο που έχει επικαλεστεί ο πρόεδρος Ολόντ βεβαίως οδήγησε σε πολύ πολύ μεγάλη σύγχυση. Σύγχυση και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Στην αρχή έπρεπε να ψάξουν να βρουν τι είναι αυτό το άρθρο, δεν υπήρχε καμία προετοιμασία για το τι κάνουμε και πώς ε, προχωράει αυτή η διαδικασία. Τι να σας πω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ σας λέω, κανείς δεν ήξερε ακριβώς τι περί πρόκειται, έτσι, κανείς. Και το λέμε και στην έκθεση. Είναι πολύ δύσκολο. Και αν θέλετε, υπάρχει και το 222 ένα άρθρο που περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες, αν θέλετε, προτάσεις για τη συνεργασία με τα κρατημέλη. Εν πάση περιπτώσει, με τη σημερινή κατάσταση ως έχει, όλα αυτά θα πρέπει να τα εκφράσουμε με μεγάλη προσοχή. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια, είπα κάποια πράγματα και θα επαναλάβω κάποια από αυτά το θέμα του Σέγγεν, οι συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα σε πολλά κράτη-μέλη, το κλείσιμο των συνόρων, η αποτυχία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέντε κράτη-μέλη, αν θέλετε, πέντε, πέντε κράτη-μέλη μόνο, αν θέλετε, στέλνουν τα συγκεκριμένα στοιχεία που τους ζητείτε στην Europol. Πέντε μόνο. Και όχι οι μεγάλες. Καμία μεγάλη χώρα, ούτε δική μου. Και το ίδιο ακριβώ γίνεται και με την Frontex, το ίδιο ακριβώ γίνεται και με την Eurojust. Έχουμε αυτούς τους οργανωμένους φορείς για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Δεν θα ήταν λογικό να συνεργαστούμε μαζί τη. Και να μην λέμε μετά απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, απέτυχε το εγχείρημα. Ενώ εμεί οι ίδιοι το σαμποτάρουμε. Και όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε και νομίζω ότι βεβαίως η έκθεσή μας συμπεριλαμβάνει πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την επικαιρότητα και θα συνεχίσουμε να την επεξεργαζόμαστε βάσει αυτών των στοιχείων. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ψηφίσουμε ο σκιώδης ηγητής, ο κ. Βιαντόφσκι. Α, ξέχασα κάτι, λέει ο κ. Μπροκ. Συγγνώμη. Ξέχασα κάτι. Και νομίζω μπορώ να το αναφέρω. Η σχέση με τα κράτη. Η Μερσέντες μίλησε για τα εθνικά κοινοβούλια. Εγώ όμως θα ήθελα να πω ότι εμείς έχουμε ένα σημείο που έχει σχέση και με την έκθεση του Σφεν Γίγκολτ. Μιλάμε για τις εθνικές κυβερνήσεις και μιλάμε και για την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή τις περιφέρειες, τις κοινότητες. Πρόκειται για αρχές που όπως ξέρετε θα πρέπει να τις δεχτούμε όπως τις ορίζουν για εθνικέ νομοθεσίε. Δεν μπορούμε εμείς να υλοποιήσουμε πρότυπα τα οποία δεν υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Και εδώ βεβαίω η συνθήκη της Λισαβόνας περιέχει κάποια στοιχεία τα οποία ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί για αυτό το λόγο. Διαδικαστικό. I think... Ε, Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να συζητήσουμε για την έκθεση αυτή τώρα. Δεν έχουμε πια χρόνο και γι' αυτό ίσως να αναβάλουμε τη συζήτηση παρακαλώ. Δεν υπάρχει καν πλήρη συμφωνία ανάμεσα στους εισηγητές και εγώ θα ήθελα να προσπαθήσω να εκφραστώ και πάνω σε αυτή τη διαφορά αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Κοιτάξτε, Μπάρμπαρα, διακόπτουμε για πέντε λεπτά μόνο. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αμέσως μετά γιατί αλλιώς πράγματι δεν θα υπήρχε χρόνο. Έχουμε άλλα τρία λεπτά. Ένας ακόμα σκιώδης θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ε, ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και περιμένω να βρω την τελική της μορφή, όπως είπε και η κυρία Σπινέλη. Θα ήθελα να ζητήσω όμως από τους συζητητές το εξής. Θα ήθελα τις απόψεις σας σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλευτικών σωμάτων στην νομοθετική διαδικασία. Την ενίσχυση των διαδικασιών κίτρινης και κόκκινης κάρτας. Πιστεύετε εσείς ότι στα πλαίσια των συνθήκων και σαν τμήμα των ορθών πρακτικών μπορούμε να υιοθετήσουμε λύσεις ενίσχυσης των κοινοβουλίων. Μπορούμε να υιοθετήσουμε σαν παράδειγμα μηχανισμούς σύμφωνα με τους οποίους αν ένα εθνικό κοινοβούλιο είναι κατά μια συγκεκριμένη νομοθετική πρότασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διακόψει την νομοθετική πορεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διευκολύνει και τις διαπραγματεύσεις με τους Βρετανούς και ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε με άμεσο τρόπο ε, τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Ξέρω ότι περιμένετε τροπολογίες από τα κοινοβούλια των κρατών μελών, αλλά θα ήθελα να μου πείτε και τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια της συνθήκης. Καλώς θα ψηφίσουμε τώρα. Ελέξτε παρακαλώ αν ε, λειτουργούν ε, τα μηχανάκια καταμέτρησης. Um, I understand some colleagues don't want to check, so. No, they are doing. Uh, 18, it's okay, we can start. Nobody is too much, nobody is political group, okay. Okay, so we can start the, development. Μπορούμε αρχίσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία και θα αρχίσουμε με την γνωμοδότηση που ετοίμασε η Mercedes Bresso, τροπολογία πρώτη υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 5 υπέρ, κατά, 4. Η τέταρτη. Δεν έκανα την τέσσερα. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 7 ε, εκτός θέματος υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 8 υπέρ κατά αποχές Μπορούμε να ελέγξουμε για την ε, τροπολογία 8, διότι το ΕΛΚ δεν ψήφισε νομίζω. Πέρα της ψηφοφορίας. είναι αστείο να βλέπει κανείς τι συμβαίνει. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Α, δεν λειτουργεί το δικό σας. Το μπλοκάρατε εσείς. Το βάλατε σωστά την κάρτα. Λειτουργεί τώρα. Βγάλετε τη κάρτα. Πολύ καλά. Τώρα είναι η 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά εγκρίθηκε συμβιβασμός α υπέρ εγκρίθηκε 16 υπέρ κατά υπέρ εγκρίθηκε 17 υπέρ κατά ελέγχουμε για την τροπολογία 17 άρχεται η ψηφοφορία <laughs> Closed. And it is adopted. Εγκρίθηκε. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 21 σε δύο ε, τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ θα ελέγξουμε για το τμήμα 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 24 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 25 υπέρ, κατά, ελέγχουμε για την 25. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. 26 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε για την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. 26 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 28 υπάρχει προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας, όχι. Όχι, είναι μόνο. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας, κατά, Αποχέσα. απορρίφθηκε και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Είναι μια γνωμοδότηση. Δεν είναι ονομαστική, είναι ε, ηλεκτρονική 19 και 2 αποχές. Συγχαρητήρια, η γνωμοδότηση εγκρίθηκε. Δεύτερη ψηφοφορία για την ομάδα τη διαπραγματευτική για τις διαπραγματεύσεις για το δικαίωμα έρευνας. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα αρχίσει σύντομα, αλλά φαίνεται ότι πλησιάζουμε, γι' αυτό καλύτερα να έχουμε ήδη την ομάδα έτοιμη για διαπραγμάτευση. Θυμάστε ότι είναι το ψήφισμα που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2014 από το Κοινοβούλιο και είχαμε και δύο έγγραφα εργασίας. Ψηφίσαμε για το δεύτερο έγγραφο εργασίας που ετοίμασε ο Ραμόν Χαουρέγγι στις 19 Νοεμβρίου. Έχουμε λοιπόν τα δύο αυτά έγγραφα, τις δύο αυτές κατευθύνσεις προς ανατολισμούς για την διαπραγμάτευση. Ε, η σύνθεση, ο πρόεδρος προεδρεύει, είναι κάτι συνεισμένο, Ραμόν Χουαρέγγι, εισηγητής και οι σκιώδες Ραγναβίλαν, Έλκα, Ραζάσκι, Σιάρμα και Πακαζάου, τον Λουάρ, της Άλντε, Χαλμουτ Σόλτς για την Κούε, Μαξ Άντερσον για τους Πράσινους, Ιζαμπέλα Αρνόλφη, Αραντιντή ε, και για ΙΕΝΕΠ. Θα πρέπει να εγκρίνουμε ηλεκτρονικά αν υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχουν ερωτήσεις, ψηφίζουμε. Αρχή, ναι, α, α, ένα λεπτό. Πέρα. Έχει πάντα προβλήματα. Έχουμε ομόφωνη αποδοχή. Είκοσι ένα Τώρα περνάμε στην, ε, στη συζήτηση πρέσσα Μπράουκ ε, εισήγηση. Σας δίνω το λόγο. Σαρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εγώ αυτό που είχα πει είναι ότι θα ήταν καλό οι δύο αυτοί οι συγητές να συμφωνήσουν, να προετοιμάσουν ένα σχέδιο ψηφίσματος. Δεν ξέρω, νομίζω έφτασα λίγο αργά, άξω όμως τον Έλμαρ Μπρόκ. Συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε. Όσον αφορά τους φιλελεύθερους, βεβαίως θα σας υπενθυμίσω κάποιες κοινοτυπίες. Πολλές φορές όμως είναι απαραίτητες οι κοινοτυπίες για να έχουμε συνοχή μου φαίνεται λοιπόν προφανές ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να λάβει υπόψη της σαφώς τις αρμοδιότητές μας, αυτές που ορίζουν οι συνθήκες. Το είπε εξάλλου ο Έλμαρ Μπροκ. Δεν άκουσα την εισηγήτρια, δεν ξέρω μπορεί να το είπατε κι εσείς. Λυπάμαι. Είναι σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες, ποια είναι τα όρια θεωρητικά τουλάχιστον ε, των συνθήκων. Εκεί που υπάρχουν δυνατότητες γιατί υπάρχουν αποτυχίες και αδιέξοδα. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά και από νομική αλλά και από πολιτική απόψεως. Για ποιου λόγους σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δράσει. Γιατί. Εν ώψη των ε, προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα για την εσωτερική ασφάλεια των χωρών μας, ο Έλμαρ μας υπενθύμησε ότι η Γαλλία αναφέρθηκε στο άρθρο, επικαλέστηκε άρθρο 47.2 και το 222 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση, τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα είδος άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για τις ε, απειλές ε, οι οποίες είναι ασύμετρες απειλές, όπως λέμε το 42.7 που αφορά με το Κάουζος Μπέλι, είναι ουσιαστικά το άρθρο 5 της αναθεωρημένης σύμβασης των Βρυξελών, που ισχύει από το 1954 για τον ΝΑΤΟ. Τώρα, το θέμα της προστασίας του θεσμικού πλασίου, του ενιαίου θεσμικού πλαισίου οι συνθήκες βεβαίως θέλουν να διατηρηθεί, να προστατευτεί αυτό το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Και για ποιο λόγο θα δημιουργήσουμε ελπίδες οι οποίες δεν μπορούν να εκπληρωθούν. Συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πολύ φοβάμαι ότι αυτά δεν υλοποιούνται σε αρκετό βαθμό. Λυπάμαι. Δεν υπάρχει όμως πολιτική όθηση και ενίσχυση για να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Τι κάνουμε, συναντιόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις για κάποια θέματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής. Συμπεράσματα όμως δεν υπάρχουν. Ανταλλάσσουμε απόψεις, αντιπαραθέτουμε απόψεις θεωρητικού αν θέλετε, περιεχομένου και ενδεχομένως μπορεί να πει κανείς ότι πρόκειται και για φλιαρία. Θα πρέπει λοιπόν σίγουρα να δώσουμε μια πολιτική χρειά σε αυτήν την έκθεση. Και παρόλες τις αντιναμίες της υπάρχουσας συνθήκης, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικά. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά και πιο αποτελεσματικά τις δυνατότητες που μας δίνει η παρούσα συνθήκη. Οι κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει σαφώς να ενισχύσουν την μεταξύ μων συνεργασία. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση λείπει η Ένωση και η Ευρώπη. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία και ελπίζω να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μου το τελικό σχέδιο έκθεσης που θα υποβάλουν οι εισηγητές. Η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ Ντανούτα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Ξεκίνησαν την εργασία τους. Εγώ θεωρώ ότι είναι μία αρχή. Εκεί βρισκόμαστε Είναι θετικές κάποιες από τις προτάσεις και είναι θετική η υπενθύμηση της κοινοτική μεθόδου και η έκκληση για την επιστροφή της κοινοτική μεθόδου σε ορισμένου τομείς. Υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς οι οποίοι θα πρέπει ακόμα να διευκρινιστούν καλύτερα. Θα ήθελα λοιπόν ανάμεσα σε εσά τους δύο εισηγητές να ζητήσω να υπάρξει μια σύμπτωση απόψεων σε τομείς τους οποίους θεωρώ σημαντικούς όπως ο ρόλος των κοινοβουλίων των κρατών μελών και η δυνατότητα χρήσης και της πράσινης κάρτας. Κατανοώ αυτό το οποίο λέγει ο Έλμαρ, ότι κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στις συνθήκες. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί η Μερσέντες να προτείνει κάτι θεωρώντας ότι οι συνθήκες μπορούν να αγνοηθούν. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν είναι ένας από τα θεματοφύλακα της συνθήκης και ένας που δεν είναι. Λοιπόν, να περάσω τώρα σε επιμέρους θέματα. Ελπίζω να εκφραστώ σωστά. Ορισμένες από τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί στα πλαίσια μιας κατεπίγουσας συγκυρίας όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σε ορισμένες χώρες έχει ουσιαστικά υπάρξει κήρυξη πολέμου. Ε, ένα άλλο θέμα κατεπήγων είναι το θέμα των προσφύγων, το θέμα των μεταναστών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, στα πλαίσια αυξανόμενων ανησυχιών στο τομέα της ασφάλειας, βλέπω να δημιουργούνται και να ακολουθούνται ε, κάποιες πολιτικές μέσα στη συνθήκη, όταν η ίδια η συνθήκη δεν δημιουργεί τον χώρο για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ έχω μία αντίρρηση αν θέλετε επί της ουσίας πάνω σε αυτό και σε σχέση με την επιστροφή στην κοινοτική μέθοδο. Ε, δεν συμφωνώ το fiscal compact να ενταχθεί ας πούμε στη συνθήκη. Δεν είναι κάτι το οποίο λειτουργήσε εκτός της συνθήκης και προφανώς και δεν θα λειτουργήσει καλύτερα εφόσον γίνει οργανικό του τμήμα, οργανικό της τμήμα της συνθήκης. Γι' αυτό λοιπόν εδώ η κάλυψη θεσμική δεν είναι κάτι το οποίο μου αρκεί. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ Γκίγκολντ. Ξεκινώντας να σας ευχαριστήσω για το κείμενο εργασίας σας. Ελπίζω η συζήτηση να είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα και επανέρχομαι εδώ στην πρώτη μου παρατήρηση. Θα πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι για την εμβέλεια της έκθεσης αυτής. Τι είναι μέσα σε αυτή την έκθεση και τι δεν είναι. Από τη μία έχουμε να κάνουμε με το θεσμικό στοιχείο, από την άλλη έχουμε να κάνουμε με το πολιτικό στοιχείο. Και σε επίπεδο πολιτικό τα πράγματα φαίνονται λίγο επιλεκτικά. Κάποιοι πολιτικοί τομεί καλύπτονται γιατί θεωρούνται σημαντικοί, κάποιοι άλλοι όχι. Αυτή είναι μια επιλογή η οποία δεν είναι προφανής απριόρι. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε απορίες. Ένα παράδειγμα. Καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Αναφέρεται. Αλλά κάποιοι άλλοι τομείς ε, οικονομικών πολιτικών δεν αναφέρονται. Δεν υπάρχει λοιπόν μια σαφής ε, διάκριση, δεν υπάρχει αν θέλετε η απαιτούμενη αυστηρότητα στις επιλογές. Το θέμα δεν είναι να καταστήσουμε σε επίπεδο πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελκυστική. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό θα λύσουμε τα θεσμικά προβλήματα που υπάρχουν και ως προς αυτό δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι συζητήσεις γύρω από τις νομισματικές και τις οικονομικές πολιτικές είναι ενδιαφέρουσες. Είναι ενδιαφέρουσες γιατί υπάρχουν θεσμικές ανησυχίες και αδυναμίες οι οποίες εκκρεμούν. Είδαμε τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει η κοινοτική μέθοδος. Νομίζω ότι καθορίζονται εδώ πάρα πολύ σωστά το τι μπορεί να γίνει σε θεσμικό επίπεδο. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε. Καταρχάς, λόγω ακριβώς της έλλειψης ε, κοινών δημοσιονομικών πολιτικών και φορολογικών πολιτικών, στα πλαίσια κοινών τμήματων της οικονομικής πολιτικής βλέπουμε την αύξηση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία στην αρχή θα ήταν ο ανεξάρτητος κυρίαρχος πολιτικός παίκτη του νομισματικού τομέα, δεν υφίσταται πλήρη πολιτικό έλεγχο και de facto έχουν καταστεί αρμόδιοι της Κεντρικής Τράπεζας για μια ολόκληρη σειρά από οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ το τι νομιμοποιούνται να κάνουν ως ανεξάρτητος εταίρος. Συνεπώς λοιπόν η ίδια η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, καθίσταται επικίνδυνη. Το να υπάρχει μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα είναι ξεκάθαρα ωφέλιμο και θεμελιώδες για μια σωστή οικονομική πολιτική. Όταν όμως βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποκτά περισσότερες εξουσίες, να διαχειρίζεται την οικονομία των κρατών που έχουν κρίση, να, να ισορροπούν τα προβλήματα της αγοράς από πλευράς επιχειρηματικότητας και μόνο, το να διασφαλίζουν τη συστημική σταθερότητα πέραν της νομισματικής αρμοδιότητας. Όλα αυτά θέτουν επιμέρους προβλήματα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στη συνθήκη. Γι' αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ένα δεύτερο θέμα είναι ο ρόλος του Eurogroup. Η έκθεση προτείνει να υπάρχει ε, μια, ένας μόνιμος δημοκρατικό υπόλογος πρόεδρος του Eurogroup. Καλή ιδέα. Απ' την άλλη όμως δεν λύνει τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με το ίδιο το Eurogroup. Ένα σώμα το οποίο είναι τόσο ισχυρό, ένα σώμα το οποίο δεν έχει ούτε καν ε, κανονισμό λειτουργίας, δεν κρατάει καν πρακτικά και όλες οι συζητήσεις του είναι ανεπίσημες. Ένα τόσο σημαντικό σώμα είναι προβληματικό και οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες οι οποίες ε, οδηγούν στο Συμβούλιο δεν είναι όσο διαφανείς όσο θα έπρεπε να είναι και όσο είναι άλλες διαδικασίες διαφανής στην Επιτροπή σαν παράδειγμα. Θέματα λοιπόν τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, το θέμα των εξωτερικών συνόρων, το θέμα της μετανάστευσης δηλαδή. Εμείς ε, είμαστε ικανοποιημένοι που προτείνονται ορισμένα μέτρα για τα θέματα της πολιτικής μετανάστευσης και χορήγησης ασύλου θα θέλαμε όμως να υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για την κατανομή ε, των ανθρώπων αυτών, των προσφύγων ανάμεσα στα κράτη-μέλη όταν ζητούν προστασία. Αυτό το οποίο χρειαζόμεθα αν θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτά τα εσωτερικά μας σύνορα. Από την άλλη υπάρχει η σαφής έλλειψη εδώ μιας πλήρους αναφοράς στο ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει όπου να είναι τελειώνω έλμα. Όχι Έλμα Χερμπρόκ, συγγνώμη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ελείπει μια σαφής ανάληψη υποχρέωσης προστασίας των δικαιωμάτων. Ακολουθεί πολιτικές οι οποίες εν μέρη ή ακροφυγώς αναφέρονται, δεν μπορεί να δημιουργεί διαδικασίες και κανόνες οι οποίες θα αποτρέπουν και θα αποκλείουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ, ο Καστάλντο έχει το λόγο. Καστάλντο δεν θες... Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία Φάμπιο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές, οπότε θα δώσω τώρα πια το λόγο στους δύο εισηγητές. Να υπάρχει ο ορισμός για το ποιό θα μιλήσει πρώτο και ποιος θα μιλήσει δεύτερο. Θα κάνουμε το ίδιο. Τώρα θα μιλήσω εγώ πρώτο. Λοιπόν, οι συνθήκε είναι ξεκάθαρε, Πολύ ξεκάθαρε. Υπάρχει το κίτρινη κάρτα. Η Επιτροπή πρέπει να αιτιολογήσει γιατί κτλ. κτλ. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα οι μισές χώρες χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής να αν θέλετε ε, μην εφαρμοστεί μια νομοθεσία ή να διακοπεί η διαδικασία για ένα νομοθετικό κείμενο και αυτό μπορεί να το κάνει είτε το Συμβούλιο είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το 55% των Εθνικών Κοινοβουλίων υπάρχει δυνατότητα μία νομοθετική πρόταση για λόγους είτε αναλογικότητας είτε επικουρικότητας μόνο για αυτούς τους δύο λόγους να απορριφθεί και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι υποχρεωμένο το Συμβούλιο πρέπει να διακόψει αυτή τη διαδικασία την νομοθετική. Αλλά επαναλαμβάνω χρειάζεται 55% των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ωραία, αυτή είναι η ιδέα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων προφανώς που θα λάβουν χώρα με την ε, Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό βασίζεται στις δυνατότητες που δίνει η παρούσα συνθήκη. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα λογικό αποτέλεσμα και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ποιε είναι οι θέσει των ΜΕΝ και των ΔΕ και όχι μόνο της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι λογικό για όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια αυτό. Το θέμα της αναλογικότητας και της επικουρικότητας είναι κάτι που σε κάθε περίπτωση και για τις πράσινες κάρτες αλλά και για άλλους που έχουν θίξει το θέμα αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί. Είναι θετικό αλλά χρησιμοποιείται για λάθος σκοπούς και έχει αρνητικές συνέπειες καταχρηστική είναι η διαδικασία. Θέλουμε λοιπόν εδώ βεβαίως να δούμε ποιος έχει την πρωτοβουλία, τα εθνικά κοινοβούλια. Επαναλαμβάνω όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Το θέμα είναι να υπάρχει πρωτοβουλία και με την δική του, αν θέλετε, πλειοψηφία, το κάθε Ευρωπαϊκό ε, Εθνικό συγγνώμη, Κοινοβούλιο των Ευρωπαϊκών Χωρών μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Τώρα, η πορτοκαλή κάρτα δεν χρησιμοποιείται από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και πρέπει να συζητήσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε αν με αυτές τις 8 εβδομάδες και πολύ εγκαίρος και αφού μεταφραστούν τα κείμενα σε όλες τις γλώσσες, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχει μεταφραστεί το κείμενο, έτσι ώστε να δοθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο και να προλάβει σε μια φάση προετοιμασίας, πριν δηλαδή αποφασιστεί και ψηφιστεί το τελικό κείμενο, να ασχοληθεί με αυτό το κείμενο. Αλλά επαναλαμβάνω πρόκειται για κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας με την προβλεπόμενη προθεσμία 8 εβδομάδων. 8 εβδομάδες χρειάζονται. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει κάπως να απλοποιηθεί έτσι ώστε να βρεθεί ένας τρόπος δεν ξέρω τώρα ποιε θα είναι οι απλοποίησει και οι ελαφρύνσεις, αλλά ε, σίγουρα αυτή η διαδικασία πρέπει κάπω να αλλάξει και να γίνει λίγο πιο λειτουργική και αποτελεσματική από ό,τι γίνεται σήμερα. Τα όρια τώρα της συνθήκης είπατε. Ναι, εννοώ ότι αυτό πρέπει να γίνει αν θέλετε τηρώντας βεβαίως τα όρια και τους περιορισμούς της συνθήκης με έναν λίγο διασταλτικό τρόπο, έτσι το κατανοώ εγώ. Και το 42.7, το πρώην 22 άρθρο, που φυσικά αφορά την πρόσφατη, αν θέλετε, κατάσταση στην Ευρώπη, το 42.7 προβλέπει τον συντονιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως ποιος συντονίζει. Ωραία, στέλνουμε δυνάμεις. Ποιος συντονίζει. Οι Αμερικάνοι. Καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι καθοριστικό αυτό ο συντονιστικός ρόλος. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, σώνουμε ζωές και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο, αν έχουμε αυτή την προληπτική δράση, δαπανώνται και λιγότερα κονδύλια, γίνεται εξοικονόμηση. Κυρία Σπινέλη, θέσατε μία ερώτημα και είπατε τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία. Ε, ε, ε, τι να σας πω. Είναι απλό. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τα πράγματα είναι απλά, δεν ενσωματώνονται κάποια πράγματα στο κείμενο της έκθεσης. Κανείς δεν μπορεί να είναι 100% ικανοποιημένος. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Πράσινη κάρτα απάντησα. Σίγουρα θα βρούμε έναν τρόπο μέχρι το Στρασβούργο να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Το Fiscal Pact, Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια πρόταση που εδώ και πέντε χρόνια, εδώ και πέντε χρόνια ακούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στην συνθήκη. Η Μεγάλη Βρετανία θέλει κάποιες εγγύησεις ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την ενιαία ώρα. Είναι λογική η απέτησή της, η ανησυχία της. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε κάθε περίπτωση αυτό το fiscal pact φυσικά θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί με τις ε, αρμοδιότητες που απορρέουν. 27, 27 χώρες από τις 28 το έχουν κυρώσει. 27 από τις 28. Μην το ξεχνάμε αυτό. Κύριε Γκίγκολτ. Μιλήσατε για το θεσμικό ή το πολιτικό. Κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν με θεσμικό τρόπο. Αλλά όχι αυτά που είναι πολιτικά. Και φυσικά είναι σημαντικό όταν πρόκειται για πολιτικά θέματα να σιγουρεύουμε και να εξασφαλίζουμε ότι λύνονται λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική τους πτυχή. Και ο καθένας βεβαίως προσπαθεί να βάλει τις πολιτικές του προτεραιότητες. Για όλους αυτούς τους λόγους επαναλαμβάνω ότι θα παραμείνουμε στα όρια τα οποία το θέμα τώρα των προσφύγων. Ναι, βέβαια, μπορούσαμε να κάνουμε πολύ παραπάνω. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε αυτή την έκθεση όλο το θέμα το προσφυγικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα και άλλα θέματα με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν επιτήρηση του τραπεζικού συστήματος, παραδείγματο χάρη, ο ρόλος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευτυχώς όμως ε, ακόμα επικρατούν ευρωπαϊκές λύσεις. Θέμα της διαφάνειας. Να βρεθούν λύσεις για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Εδώ προτείνουμε όμως αν θέλετε, ο υπεύθυνος, ο αρμόδιος για την οικονομική πολιτική επίτροπος, ο οποίος βεβαίως είναι αρμόδιος και για όλα όσα συμβαίνουν στην Ευρωζώνη, να έχει αρμοδιότητα και για το Eurogroup. Αυτό θα ήταν μια λύση. We are ε, already beyond the time for the ε, very... Έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις γρήγορες υποχρεωτικά παρατήρησεις τους. Από τον Έλμαρ μπορούμε να καθορίσουμε μια συνάντηση με τους συντονιστές, τους σκιώδεις μάλλον, για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Θα δούμε αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, όχι πάνω σε αυτό το κείμενο, αλλά πάνω στο τελικό επίσημο. Το θέμα των κοινοβουλίων των κρατών μελών είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολύ. Είναι προφανές ότι το θέμα το οποίο τίθεται δεν αφορά στη διαχείριση της επικουρικότητας, επί της οποίας υπάρχουν πρωτοβουλίες και για το αν θα υπάρξει μια κόκκινη κάρτα που θα μοιάζει πολύ με την πορτοκαλί που δεν χρησιμοποιείται. Το αίτημα είναι να υπάρξει μια μεγαλύτερη δυνατότητα συνεργασίας δύο θα έλεγα κατευθύνσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει την ίδιο, το ίδιο τη δυνατότητα πρωτοβουλίας, αλλά μπορεί να συντάξει εκθέσεις πρωτοβουλίας. Αν περιοριστεί σε αυτό, οι προτάσεις του είναι απόλυτα νομιμοποιημένες, γιατί ε, στα πλαίσια μιας πρότασης ε, που λέγεται πράσινη κάρτα, τα εθνικά κοινοβούλια πήραν κάποιες αποφάσεις εισαγωγικά σχετικά με την COP21 και κανένας δεν τους είπε ότι δεν έπρεπε να το κάνουν. Υπάρχει λοιπόν μια πρωτοβουλία επιμέρους περιορισμένη νομοθετική την οποία έχει το Κοινοβούλιο. Τώρα οι συνθήκες προβλέπουν μια διοργανική συμφωνία που λέγει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να λάβει υπόψη τις προτάσεις αυτές. Μέχρι εδώ παραμένουμε στο εσωτερικό των συνθήκων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε από κοινού εάν έχει ενδιαφέρον οι προτάσεις αυτές να θεωρηθούν σαν μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Τώρα, για να υπάρξουν μέσα διακανονισμένα και εφαρμόσιμα με δεσμευτικό τρόπο, τότε θα απαιτηθούν τροποποιήσεις στις συνθήκες, οπότε τότε μιλάμε για την έκθεση Φερχόστατς γύρω από μια σειρά άλλων θεμάτων σημαντικών που, έφεσαν, που έφεσε η συνάδελφος κυρία Σπινέλη. Πράγματι πιστεύω ότι ε, εδώ υπάρχει το επαρκές επίπεδο τεκμηρίωσης και το λέω αυτό και για τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Σβεν Γίγκολντ. Όλο το κομμάτι της ζώνης ευρώ είναι κάτι το οποίο απαιτεί την επιστροφή σε κοινοτική μέθοδο παρά τις περιπλοκότητες που υπάρχουν στο εσωτερικό της συνθήκης και οι οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω τροποποίησής της. Τώρα, για το ε, δημοσιονομικό σύμφωνο, είναι κάτι το οποίο βγαίνει από τη δική μας αρμοδιότητα. Έτσι και αλλιώς απαιτείται να υπάρξει ένταξη στη συνθήκη, οπότε τροποποίηση υποχρεωτικά της συνθήκης. Και όποιος μιλάει τροποποίηση της συνθήκης, μιλάει για αλλαγή της συνθήκης που έχει υπογραφεί από τις χώρες και της ζώνης ευρώ και τις άλλες. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο διαφεύγει θα έλεγα της δικής μας εκθέσεως και τίποτα δεν αποκλείεται ότι αν δεν υπάρξουν προτάσεις λειτουργικές από πλευράς μας να υπάρξει μια νέα συνθήκη συμπεριληφθούν αυτές οι προτάσεις σε μια νέα συνθήκη. Τώρα για τις υπερβολικές αρμοδιότητες και εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό δείχνει ότι στο εσωτερικό της συνθήκης υπάρχει περιθώριο να γίνουν. Γιατί έτσι κι αλλιώς 10 συνταγματολόγοι θα διαβάσουν με 10 διαφορετικούς τρόπους τη συνθήκη αλλά βασικό στόχος της δικής μας πρότασης είναι να αποστείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο να λέγει ότι στο εσωτερικό της συνθήκης μπορεί κανείς να επιστρέψει στη λεγόμενη κοινοτική μέθοδο αλλά και να ενισχύσει τη συγκεκριμένη μέθοδο και από την άλλη μπορούν πάρα πολλά να γίνουν στο τομέα της οικονομίας, της άμυνας, της ασφάλειας και των κοινωνικών θεμάτων θέματα πάνω στα οποία από πλευρά των κρατών μελών, από πλευρά των πολιτών, από πλευρά των ευρωβουλευτών, από πλευρά των βουλευτών των Εθνικών Κοινοβουλίων, συνεχώς καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πράγματα και να τα κάνει με ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τη συνθήκη όπως ακριβώς το κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέναντι στη μεγάλη οικονομική κρίση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ελπίζουμε η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας να γίνει στα μέσα Μαρτίου. Οι επιλογές είναι ανοιχτές όμως και οι δύο εισηγητές είναι διαθέσιμοι. Αν κάποιος έχει γραπτά σχόλια και θέλει να συνεισφέρει θα τα δεχτούν. Αλλά οι τροπολογίες οι πραγματικές θα γίνουν στην τελική πρόταση. Λοιπόν, στις 3 θα συνεχίσουμε ακριβώς για την επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ, τελειώσαμε.